Nous allons maintenant aborder Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Με το θέμα αυτό ξαναγυρνάμε στις συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είχαμε κληρονομήσει από την προηγούμενη κοινοβουλευτική εντολή. Η πρώτη συζήτηση, όπως αποφάσισαν οι συντονιστές, αφορά την κατάσταση των συνδικάτων στην Κολομβία. Επιτρέψτε μου λοιπόν να καλωσορίσω όχι μόνο τους ομιλητές μας, αλλά και τα μέλη άλλων ενδιαφερομένων κοινοβουλευτικών επιτροπών, της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου, των Εξωτερικών Υποθέσεων και των μελών της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να καλωσορίσω επίσης τον κύριο Σάλα Φράγκα, πρόεδρο της ε, διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη διακοινοβουλευτική συνέλευση Eurolat να καλωσορίσω επίσης όλος ιδιαιτέρως στον Υφυπουργό Εργασίας της Κολομβίας, τον κύριο ε, Ρικάντρο Ανδρές Ετσεβερία Λόπες. Εκπροσωπεί την Κολομβιανή κυβέρνηση και συνοδεύεται από τον πρέσβη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση έχει στενές σχέσεις με την Κολομβία και είναι φυσιολογικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητά προσεκτικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόσφατα πήραμε πληροφορίες για έναν πολλαπλασιασμό των επιθέσεων εις βάρος των σονδικαλιστών και ένα εχθρικό κλίμα προς τους εργαζομένους που προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Οι πληροφορίες που πήραμε πολλές φορές είναι αντιφατικές και ελπίζουμε ότι η συζήτηση αυτή να μας επιτρέψει να δούμε καλύτερα τα πράγματα. Η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου προβλέπει μια ανταλλαγή απόψεων για την Κολομβία την Τετάρτη που να έχει σαν στόχο τις υποχρεώσεις που προέρχονται από το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων. Όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει ξεκινήσει μια ζωηρή συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις τις οποίες διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία Ελευθέρωσης των Αλλαγών με την Κολομβία. Λόγω του πεδίου δράσης της Επιτροπής μας, οι σημερινές συζητήσεις θα έχουν σαν στόχο την σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Κολομβία την χάνει βοήθειας μέσα από το Ταμείο Βοήθειας για την Ανάπτυξη και θα πάρει 160 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Είναι λοιπόν δική μας ευθύνη να ασχοληθούμε με τον τρόπο με τον οποίο συνοδεύεται αυτή η βοήθεια από τον διάλογο για την στήριξη των ανθρωπίνων των δικαιωμάτων. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στον κύριο Μίτσελ. Ο κύριος Μίτσελ θα κάνει εισαγωγή στο θέμα πριν ακούσουμε τις απόψει των υπολείπων ομιλητών. Κύριε Μίτσελ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Thank um, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι η πρώτη ακρόαση που ε, διοργανώνει η Επιτροπή μας και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων στην Κολομβία και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων στην Κολομβία. Αναφερθήκατε στα 160 εκατομμύρια που προβλέπονται για την περίοδο 2007-2013. 32 εκατομμύρια έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ο κύριος Βάνεγκας είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ε, μεγαλύτερης νομοσπονδίας ε, συνδικαλιστικής της Κολομβίας, της CUT, Colombian Trade Union Congress, Επίσης έχουμε μαζί μας την κυρία Ντούμπια Ονρή που είναι διευθύντρια των Διεθνών Εργασιακών Προδιαγραφών του, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και έχουμε επίσης μαζί μας τον κύριο Κάρλος Χόλμες Τρίλο Γκαρθία, ο οποίος είναι πρεσβευτής της Κολομβίας, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κάνω κάποιε εισαγωγικέ παρατηρήσει. Όπω ξέρουμε, η Κολομβία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ανθρωπιστική φύση και προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε εκτελέσει χωρί να έχουν προηγηθεί δίκε, μετατοπισμό πληθυσμών και πολλές φορές εσωτερικές διενέξεις που επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι Πολύ συχνά οι εργαζόμενοι γίνονται αντικείμενο επιθέσεων, απαγωγών, ε, βιοπραγιών. Η κατάσταση αυτή σαφώς είναι απαράδεκτη. Συντοπιώ από διάφορες επαφές που είχαμε με την Κολυμπιανική κυβέρνηση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι ότι μπορούν ποτέ οι εργαζόμενοι να βρίσκονται σε τόσο άσχημη, δυσάρεστη θέση μόνο και μόνο επειδή θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδικαλιστές οι οποίοι έχουν πέσει θύματα βιοπραγιών που έχουν χάσει τη ζωή, της, τη ζωή τους και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε μαζί μας τους προσκεκλημένους μας προκειμένου να μας ενημερώσουν για το πώς έχουν τα εργασιακά δικαιώματα στην Κολομβία και το τι έχει γίνει στη χώρα αυτή, αν έχει όντως αλλάξει η κατάσταση ή όχι. Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η δολοφονία συνδικαλιστών ή ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι το εντελώς απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. The... Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βάνεγκας από την Colombian Trade Union Congress, CAT. Και σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τον χρόνο μιλίας, έχετε 10 λεπτά Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απευθύνεται. Ευχαριστώ την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, για την ε, ευκαιρία που μας δώσατε να δώσουμε μια μαρτυρία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ε, συνδικαλιστών της Κολομβίας είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με την έγκριση μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Κολομβία. Η ύπαρξη αυτής της κατάστασης και αντίστοιχη συζήτηση υπήρξαν καθοριστικές για να ανασταλούν ή να μην επικυρωθούν οι συμφωνίες ελεύθερης εμπορικής σχέσης με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και ε, την ομάδα των βόρειων των χωρών. Υπό την έννοια αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την δυσμενή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις των συνδικαλιστικών ελευθεριών, όπως διαπιστώθηκε πολλές φορές από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας που στην τελευταία του συνεδρίαση ε, είπε ότι η Κολομβία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 25 χωρών με τις περισσότερες παραβιάσεις των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Η Κολομβία έχει το θλιβερό ρεκόρ του 60% συνδικαλιστών που έχουν δολοφεθεί τα τελευταία χρόνια. Ε, και κατά τη διάρκεια του 2009 δολοφονήθηκαν 40 συνδικαλιστές, το 2008 49 και το 2007 39 ε, συνδικαλιστές. Όλες αυτές οι περιπτώσεις περιβάλλονται από μια, ένα καθεστώς ατιμορρυσία παρά την ε, δήλωση της ε, κυβέρνησης ότι θέλει να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη. Η συστηματική παραβίαση της, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επιθέση κατά της σωματικής ακαιρεότητας των συνδικαλιστικών της Κολομβίας εκφράζεται από το γεγονός ότι το 2009 εκφράστηκαν πάρα πολλές απειλές κατά της ζωής των συνδικαλιστών και 44 αναγκαστικές εκτοπίσεις, 6 περιπτώσεις ε, βασανισμού κλπ. Και όλα αυτά ε, με 29% ποσοστό ατιμορρησίας. Ε, οι απειλές κατά τη ζωή των συνδικαλιστών είναι πάρα πολλέ και κάθε μέρα παρατηρούνται ε, σχεδόν παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των συνδικαλιστών της Κολομβία. Κατά τη διάρκεια του, της θητείας του Προέδρου Αλμπορία ε, δολοφονήθηκαν πάνω 500 συνδικαλιστέ. και, ε, και παρατηρήθηκαν 36% των συνολικών ανθρωποκτονιών ενώπιον των ε, διεθνών ε, οργανισμών καταγγείλαμε την ευθύνη της ε, κυβέρνησης που εκ παραλήψεως δεν μπόρεσε να εγγυηθεί τη ζωή των πολιτών της χώρας. Η, η ευθύνη αυτή στην οποία, την οποία αποτυγχάνει να αναλάβει η κυβέρνηση της Κολομβίας γιατί είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως για παράδειγμα η περίπτωση ε, Νογέρα, ο οποίος ε, ανακρίνεται γιατί παρέδωσε ένα κατάλογο ε, συνδικαλιστών στην κυβέρνηση, οι οποίοι στη συνέχεια δολοφονήθηκαν. Επίσης υπήρξε περίπτωση μιας εξοδικαστικής εκτέλεσης και υπάρχουν πολλοί στρατιωτικοί οι οποίοι εκτίουν τις ε, ποινές στη φυλακή και πολλοί ανακρίνονται. Ε, τον Ιανουάριο παραστρατιωτικοί ανακρίνονται για 1.700 εξοδικαστικές εκτελέσεις νέων σε ορισμένες περιπτώσεις συνδικαλιστών οι οποίοι ε, δολοφονήθηκαν ενώ ήταν εντελώς ε, αθώοι και οι ένοχοι δεν οδηγήθηκαν στην ε, δικαιοσύνη. Ε, με τώρα από αυτό συνεχίζεται ένα καθεστώς ατιμορρησίας όσον αφορά αυτές τις 1600 εξοδικαστικές εκτελέσεις. Και όλοι αυτοί οι αριθμοί δείχνουν μια τεράστια κρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του συνδικαλισμού όσον αφορά την ύπαρξη μιας βίας η οποία είναι διάχυτη και αδιάκριτη προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενώ η κυβέρνηση τελικά προσπαθεί να συγκαλύψει την πραγματική διάσταση του προβλήματος. Ε, πρόκειται για μια συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ε, συνδικαλιστών και θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια πολιτική, σαν μια μορφή πολιτικής γενοκτονίας κατά του συνδικαλιστικού κινήματος. Ε, έναντι αυτής της κατάστασης οι συνδικαλιστικές ενώσεις, οι οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάνω από 400 οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών στην Κολομβία ε, ελπίζουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων. Και εμείς ταχθήκαμε όλοι από κοινού κατά της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με την Κολομβία και αναγνωρίζουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν βάλει στην άκρη η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπω αυτό τη Κολομβία που συνεχίζει να δολοφονεί συνδικαλιστέ και προασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό το γεγονό το οποίο έχει αναγνωριστεί και έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη σε άλλε χώρε όπως δείχνει η ομιλία του Προέδρου της ΗΠΑ καθώς και οι προσπάθειες της γυρωσίας στον Καναδά το θέμα αυτό στις χώρες αυτές ε, τέθηκε στο επίκεντρο ούτως ώστε να παγώσουν οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Κολομβία. Μία κυβέρνηση η οποία, ε, στην οποία έχουν τεθεί τόσες ερωτήσεις ε, για ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων νομιμοποιείται εφόσον συνεχίσει το καθεστώς ε, ατιμορρησίας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να σταλούν οι συμφωνίες όσο υπάρξει ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς ζητούμε να ληφθεί σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης όσον αφορά την επικύρωση της ε, Συμφωνίας ε, Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολομβίας και θα πρέπει η Διεθνής ε, Συνομοσπονδία Συνδικάτων να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Η συνάδελφος από την ε, Συνομοσπονδία Εργαζομένων της ε, Κολομβίας θα απευθύνει ένα χαιρετισμό και θα σπεί κάποια πράγματα εν σχέση με τη θλιβερή κατάσταση των συνδικαλιστών στη χώρα αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Euh, Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Ντούμπια από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Έχετε και εσείς 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Thank uh, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να κάνει μια παρουσίαση εδώ στην συνάντησή σας. Θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στο, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Είμαστε η γραμματεία ουσιαστικά της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και ως γραμματεία της οργάνωσης αυτής θα εκφράσω τις απόψεις της οργάνωσης αυτής. Organize Convention 87 and the right to organize. Η Κολομβία έχει επικυρώσει και τις δύο συμβάσεις για τις ε, συλλογικές συμβάσεις αφενός και για, την, για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε αφετέρου. Τα όργανα επιτήρησης ε, του ILO και συγκεκριμένα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των συστάσεων καθώς επίσης και η Επιτροπή για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεστε έχουν ε, σχολιάσει πολλές φορές στο παρελθόν ήδη από, το τέλο της δεκαετίας του 1980 την εφαρμογή των συμβάσεων αυτών στην Κολομβία. Και πιο συγκεκριμένα τα όργανα αυτά έχουν εξετάσει καταγγελίες για τη χρησιμοποίηση βίας κατά των συνδικαλιστών, συγκεκριμένα χιλιά άτομα έχουν πέσει θύματα, και για την κατάσταση ατιμορρησία στην Κολομβία. Η κυβέρνηση Κολομβίας μας έχει πει ότι στην περίπλοκη κατάσταση βίας στην Κολομβία, που ουσιαστικά υποστηρίζεται κυρίως από παραστροτικές ομάδες, από αντάρτικες ομάδες, καθώς επίσης και από ομάδες διακίνησης ναρκωτικών, όλοι οι τομείς της κοινωνίας έχουν επηρεαστεί και όχι μόνο οι συνδικαλιστές. Επίσης γίνανε κάποια σχόλια όσον αφορά νομοθετικά ζητήματα. Σε ορισμένες αποστολές άμεση επαφής από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας έχουν λάβει χώρα στην Κολομβία από την δεκαετία του 90 και μετά, αλλά δεν έχει σημειωθεί κάποια ιδιαίτερη πρόοδος. Το 1998 μια καταγγελία για μη συμμόρφωση με την Σύμβαση Παριθμών 87 υπευλήθη στο Διεθνές Γραφείο, στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας από 27 αντιπροσώπους κατά της Κολομβίας. Τα αρμόδια όργανα του ΑΕΛΟ αποφάσισαν να μην δημιουργήσουν αμέσω μια ερευνητική επιτροπή και πρότειναν να γίνει μια αποστολή άμεση επαφή με του αρμοδίου Κολομβία το 2000. Μετά την αποστολή αυτή, η κυβέρνηση πήρε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επικυρωποιήσει την Σύμβαση Παριθμών 151 όσον αφορά τις εργατικές σχέσεις, καθώς επίσης και τη Σύμβαση 154 για τις συλλογικέ συμβάσεις και επίσης αποφάσισε να τροποποιήσει ή να καταργήσει ένα πολύ σημαντικό αριθμό νομοθετικών κειμένων και να δώσει τους απαραίτητους πόρους για την προστασία των επικεφαλήσεων συγκαλικών οργανώσεων και των συνδικαλιστών εν γέννη. Την εποχή εκείνη η κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει μια ειδική επιτροπή για την διαχείριση των συγκρούσεων που είχαν να κάνουν με το ζήτημα της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε. Μετά από κάποια λοιπόν χρόνια αφού έγινε μια αξιολόγηση των νέων αυτών μέτρων και ενώ είχαν διατηρηθεί ακόμα βαθιές ανησυχίες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση βίας κατά των συνδικαλιστών, ο ILO αποφάσισε να μην δημιουργήσει μια επιτροπή ερεύνας. Μεταξύ του 2000 και του 2007 ένας ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Διευθυντή του ILO, καθώς επίσης και αποστολές ε, υψηλού επίπεδου πήγανε στη χώρα. Ήδη από το 2006 υπεγράφει μία τριμερής ε, συμφωνία για την ελευθερία του ε, συνεταιρίζεσθε από εκπροσώπους κολομβιανής κυβέρνησης και από τους κοινωνικούς εταίρους στη Γενέβη. Στην συνεδρίαση του 2009 της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προδιαγραφών εξέτασε για άλλη μια φορά την εφαρμογή της Συμβάσης 87 από την Κολομβία και κάλεσε την κολομβιανή κυβέρνηση να συνεχίσει να δέχεται την υποστήριξη του ILO όσον αφορά τα κρεμή ζητήματα. Η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να ενδυναμώσουν το κοινωνικό διάλογο στην Κολομβία. Μετά την Διεθνή Διάσκεψη του 2009 του ILO, η κυβέρνηση της Κολομβίας με προσκάλεσε να επισκεφθώ την χώρα προκειμένου να δω τι πρόοδος είχε σημειωθεί με την εφαρμογή των συμβάσεων υπαριθμών 87 καθώς επίσης και ε, όσον αφορά την εφαρμογή των συμπερασμάτων της τριμερού συμφωνίας για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και τη δημοκρατία. Στα πλαίσια της εντολής της ε, αποστολής αυτής και ε, ευθυγραμμιζόμενη με τα συμπεράσματα της Επιτροπής της Διάσκεψης για την εφαρμογή των προδιαγραφών αποφασίστηκε να εντοπιστούν πληροφορίες για τα εξή τρία σημεία. Καταρχάς, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να καταπολεμηθεί η τιμωρησία και να σταματήσει η βία κατά των συνδικαλιστών. Δεύτερον, ποιε είναι όμω τα νέα νομοθετικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση και τα οποία είχε συστήνει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του ILO. Και τρίτον, να εξεταστεί πώ λειτουργούσε η Ειδική Επιτροπή για την Διαχείριση των Συγκρούσεων πριν ληφθούν οι αποφάσει του ILO. Όσον αφορά τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί η βία κατά των ε, συνδικαλιστών και όσον αφορά το ζήτημα της ατιμορρησίας, έλαβα πληροφορίες όσον αφορά νομοθετικά και άλλα μέτρα τα οποία εγκρίθηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρθηκαν σε στατιστικά δεδομένα όσον αφορά τι βιοπραγίε και όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τι βιοπραγίε κατά των συνδικαλιστών και γίνονται επίση αναφορές στις συλλήψεις και καταγγελίες ε, κατά των ε, υπευθύνων για τις πράξεις αυτές. Η προστασία των επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων αναφέρθηκε επίσης στις συναντήσεις αυτές. Επίσης ε, αναφερθήκαμε στην υπόθεση 1787 η οποία είχε συζητηθεί και στην Επιτροπή για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθε. Όσον αφορά τα νομοθετικά ζητήματα, σημείωσα συγκεκριμένα κάποιες δικαστικές αποφάσεις που αντιμετώπιζαν πολλά από τα ζητήματα που είχαν εντοπιστεί και εξέτασε και την επιρροή που θα είχαν τέτοιες αποφάσεις. Όσον αφορά την ε, λειτουργία της ε, Τριμερούς Επιτροπής, με συμμετοχή του ILO, έλαβα πληροφορίες για τη λειτουργία της Επιτροπής αυτής. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τόνισαν ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί ο ρόλος της Επιτροπής αυτής. Στο τέλος λοιπόν της αποστολής μου πρότεινα να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα τα οποία εξετάζουν τα όργανα επίβλεψης του ILO. Στο τέλος της αποστολής αυτής, η κυβέρνηση, σε μία ανακοίνωση που μου έδωσε σε μένα προσωπικά, που δόθηκε σε μένα προσωπικά, με συγχωρείτε, μέσω του Υπουργού Κοινωνικής Προστασίας. Η κυβέρνηση λοιπόν δεσμεύτηκε να εγκριθούν ακόμα περισσότερα μέτρα μετά από συστάσεις που είχε κάνει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του ILO, καθώς επίσης και μετά από συστάσεις που είχε κάνει η Επιτροπή για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε όσον αφορά τις βιοπραγίες, όσον αφορά το ζήτημα της ατιμορρησίας, όσον αφορά την προστασία των συνδικαλιστών και των επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής αυτής της τριμερούς στην οποία αναφέρθηκα, όσον αφορά τις συστάσεις της Επιτροπής του συνεταιρίζεστε και όσον αφορά τα υπόλοιπα νομοθετικά κρεμή ζητήματα τα οποία εντόπισε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και όσον αφορά το ζήτημα της τεχνικής υποστήριξης από τον ILO. Δεν θέλω να αφαιρθώ σε όλα αυτά τα ζητήματα σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί ο χρόνος ομιλίας είναι περιορισμένος. Η Επιτροπή των Υπερογνωμόνων για την εφαρμογή των συστάσεων και των συμβάσεων στις παρατηρήσεις που έκανε το 2009 και τις οποίες έδωσα στην Επιτροπή σας πριν τη συνεδρίαση αυτή. Και αυτό το έκανα αποτελεί μια εξαίρουσα αστικά στη δικασία που ακολουθούμε γιατί δεν έχουν δημοσιευθεί επίσημα ακόμα τα έγγραφα αυτά. Λέγεται λοιπόν στο έγγραφο αυτό ότι οι δεσμεύσει της κολομβιανής κυβέρνησης έχουν εκπληρωθεί και ζητάτε από την κυβέρνηση στην επόμενη έκθεσή της να αναφερθεί σε περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά τις αρχικές δεσμεύσεις. Η Επιτροπή των προγνωμόνων καταδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι περιορισμοί στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι, στο δικαίωμα της απεργίας, στο δικαίωμα των συλλογικών συμβάσεων και ότι, αυτοί, και ότι ορισμένοι περιορισμοί έχουν ε, αρθεί μέσω νέων δικαστικών αποφάσεων ή νομοθετικών μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι τα σημαντικότερα νομοθετικά εκκρεμή ζητήματα έχουν πλέον επιληθεί. Η Επιτροπή για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεστε θα εξετάσει την περίπτωση 1787 που αναφέρεται στις καταγγελίες του 1990 για την χρησιμοποίηση βίας και στη συνεδρίαση λοιπόν που θα κάνει η Επιτροπή το 2010 θα εξετάσει συγκεκριμένη αυτή περίπτωση και Ελπίζουμε ότι θα δοθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκείνης οι, τα απαραίτητα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να αποτρεπούν οι βιοπραγίες κατά των ε, συνδικαλιστών και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ατιμορρησίας. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια χωρίς ε, να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, μετά από πάρα πολλά χρόνια βίας κατά των ε, συνδικαλιστών, η κυβέρνηση μας ενημέρωσε για 218 περιπτώσεις όπου έχουν ληφθεί δικαστικές αποφάσει κατά των υπευθύνων τέτοιων βιοπραγιών. Πρέπει επίσης να πούμε ότι οι πληροφορίες που έλαβα κατά τη διάρκεια της αποστολής μου τον Οκτώβριο του 2009 δείχνουν ότι μειώνονται οι δολοφονίες των συνδικαλιστών. 196 το 2000, το 2008 και 23 δολοφονίες το 2009. Και βλέπουμε επίσης ότι οι δεσμεύσεις κυβέρνησης συμπεριλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό ποσό χρηματικό προκειμένου να προστατευτούν ακόμα περισσότερο συνδικαλιστές και προκειμένου να καταργηθεί το φαινόμενο της ατιμορρησίας, δίνοντας τους απαραίτητους πόρους προς το δικαστικό σύστημα. Εν κατακλείδη κυρία Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της τεχνικής υποστήριξής της να βοηθήσει και αυτή να καλυφθούν τα κενά τα οποία έχει εντοπίσει ο ILO. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πετύχουμε πολύ μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στον πολιτικό διάλογο και την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνεται προς την χώρα. Μολονότι έχει στην συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ILO τελευταία χρόνια, λίγε είναι οι περιπτώσει εκείνε όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια του ILO προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εφαρμογή νομοθεσία εργασιακή σε χώρε όπω η Κολομβία. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Υφυπουργού Εργασίας, τον κύριο Τσεβέρια Ιλόπες. Όπως επίσης και στον πρέσβη της Δημοκρατίας της Κολομβίας της Βρυξέλλες έχετε 10 λεπτά από κοινού παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να παρέμβω εδώ και να διευκρινίσω ορισμένα θέματα σχέση με τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι βουλευτές και ορισμένα ε, μέλη των ε, ενώσεων των εργαζομένων. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι η κυβέρνηση θλίβεται βαθύτατα για τα εγκλήματα ε, που διαπράχθηκαν στην Κολομβία εις βάρος των εργαζομένων. Αλλά σας καλώ να δούμε τους αριθμούς παρουσιάζονται εδώ σε ένα εθνικό πλαίσιο. Το 2001 στην Κολομβία δολοφανήθηκαν 27.800 πολίτες. Ένα πραγματικά, ένας αστρονομικός αριθμός που πραγματικά μας λείπει βαθύτερα. Το 2009 δολοφονήθηκαν 15.817 πολίτες πραγματικά, επίσης αστρονομικός αριθμός, αλλά που δείχνει μία μείωση της τάξης 45% της εγκληματικότητας κατά του εθνικού πληθυσμού της Κολομβίας. Το 2001 δολοφονήθηκαν 205 ε, συνδικαλιστές στην ε, Κολομβία, ένας αριθμός που πραγματικά μας θλίβει και μας ε, ντροπιάζει σε ένα διεθνές ε, πλαίσιο. Από το 2009 δολοφονήθηκαν βάσει των επίσημων στοιχείων 28 επικεφαλής των συνδικάτων. Βάσει των στοιχείων της συνδικαλιστικής σχολής 40 ε, συνδικαλιστές. Και στις δύο περιπτώσεις Εάν δούμε τα στοιχεία παρουσίασε η κυβέρνηση για αυτά που παρουσιάζει η συνδικαλιστική σχολή ε, σημειώνεται μία μείωση της τάξης του 78% εάν δούμε τα στοιχεία της συνδικαλιστικής ε, σχολής. Άρα λοιπόν η πολιτική αυτή συστηματικών δολοφονιών των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων ε, στερείται ε, βάση τα, η σύγκριση αυτών των στοιχείων, των επίσημων στοιχείων και των στοιχείων των συνδικαλιστών ε, δείχνουν ότι υπάρξει μια σημαντική μείωση ε, αυτού του αριθμού. Ε, αυτή η διαφορά έγκυται σε ζητήματα ερμηνείας. Ορισμένες ε, χρονιές ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος, ο αριθμός της συνδικαλιστικής σχολής είναι μεγαλύτερος από τα επίσημα νούμερα, ενώ άλλες ε, χρονιές ε, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Από το 2003 η επίσημη αριθμοί ήταν 101 ενώ τη συνδικαλιστική Ακαδημίας ήταν 94 ή το 2007 ο επίσημο αριθμό ήταν 26 ενώ τη συνδικαλιστική σχολή ήταν 39. Ε, βασικά βλέπουμε ότι ε, τα θύματα είναι μέλη συνδικάτων ε, και είναι ενεργά μέλη που, με κάποιες δραστηριότητε. Ωστόσο, η Συνεργαστική Ακαδημία περιλαμβάνει στα στοιχεία της και άλλα πρόσωπα εκτός των συνδικαλιστών. Δηλαδή το 12 που είναι η διαφορά για τα στοιχεία του 2009 είναι επικεφαλής του αγροτικού κινήματος που όμως δεν είναι συνδικαλιστές. Ε, προτείναμε ε, στο πλαίσιο μιας διαβούλευσης να επαναδιατεθούν τα κριτήρια τα οποία μας επιτρέπουν να ενοποιήσουμε αυτούς τους ε, δείκτες, τους στατιστικούς δείκτες. Αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε κατάλληλη μορφή διαβούλευσης. Ε, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το πράξουμε και αλλά χρειαζόμαστε γι' αυτό και την ε, συνεργασία, τη δική σας συνεργασία και την ε, συνεργασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Κολομβία, ούτως ώστε να ε, δοθεί μια σωστή εικόνα της πραγματικότητας. Αυτό το οποίο δεν δείχνουν τα στοιχεία αυτά ή που κρύβουν είναι ότι υπάρχει μια πολιτική της κυβέρνησης ε, αυτές ε, οι βιοπραγίες είναι καρπός του ένοπλου αγώνα ε, της δρομοκρατίας του ΦΑΡΚ και του ΕΛΕΝΕ και των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Στην Κολομβία δρούν τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες τρομοκρατούν τον πληθυσμό. Σήμερα έχουμε τρεις ομάδες που κινδυνεύουν. Μεταξύ αυτών είναι οι συνδικαλιστές. Αλλά Επίσης και οι δημοσιογράφοι, οι κυβερνήτες κλπ. Πριν από ένα μήνα ένας κυβερνήτης της Κολομβίας ε, κατα... σφαγιάστηκε από την ΦΑΡΚ ε, στρατιωτικοί, δήμαρχοι, βουλευτές ε, κλπ. Όλοι αυτοί πέφτουν θύματα αυτής της βίας από αυτές τις ομάδες, η ομάδα η οποία έχει μεγαλύτερη προστασία εκ μέρους του κράτους είναι οι συνδεκαλιστές. Καταρχήν υπάρχει μια, ένα τμήμα στην εισαγγελία που αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στην έρευνα, στην διερεύνηση των εγκλημάτων κατά συνδεκαλιστών. Και στο θέμα αυτό που αφορά την ατιμορρησία θα ήθελα να σας πω ότι από το 2000 μόνο, υπήρξε μόνο μία ε, καταδίκη. Ε, τώρα 69 ε, ε, καταδικαστικές αποφάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε 7, στα 7 τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αύξηση αυτών των καταδικαστικών αποφάσεων. Ε, υπάρχει όπως σας είπα ένα ειδικό τμήμα στην εισαγγελία μας αλλά υπάρχουν και ειδικοί, ειδικευμένοι δικαστές οι οποίοι είναι ειδικευμένοι να καταδικάσουν τους ενόχους υπετίους αυτών των ε, δολοφονιών, των ανθρωποκτονιών. Ε, κανένα, καμιά άλλη ομάδα του πληθυσμού που κινδυνεύει και υπάρχουν δέκα τέτοιες ευάλωτες ομάδες δεν έχει αυτής Όσον αφορά τώρα τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, από 6 εκατομμύρια δολάρια επενδύσεων το 2001 όσον αφορά το σχήμα προστασίας, περάσαμε στα 13 εκατομμύρια το δολάριο το 2009. Ε, συνεπώς η κυβέρνηση είναι, βλέπουμε ότι έχει την προφανή βούληση να προστατεύσει τους συνδικαλιστές. και επαναλαμβάνει ο μιλητή του αριθμού αυτού. Και για μια φτωχή χώρα αυτή είναι μια σημαντική επένδυση. Από τα 40 εκατομμύρια δολαρίων που επενδύονται κάθε χρόνο για την προστασία των 10 ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο, 13 ε, εκατομμύρια αφιερώνονται στην προστασία των ε, συνδικαλιστών. Συνεπώ, το να πει κανεί ότι δεν υπάρχει προστασία στην Κολομβία των συνδικαλιστών, ε, αυτή η πληροφορία είναι εντελώ παραπλανητική και είναι αντίθετη με αυτό που μας δείχνουν οι αριθμοί. Κανείς επικεφαλής του συνδικαλιστικού κινήματος που να προστατεύεται δεν έπεσε θύμα επιθέσεων κατά τη ζωή του. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει βεβαίως ένα τεράστιο πρόβλημα βία στην Κολομβία, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια έκκληση στο Κοινοβούλιο, ούτε ώστε να το αποθήσει στο σωστό πλαίσιο γιατί η βία αυτή δεν αφορά μόνο τους συνδικαλιστές, αλλά αφορά όλον τον πληθυσμό της Κολομβίας και υπάρχει ένα γενικευμένο φαινόμενο βίας. Θα ήθελα επίσης να σας πω, κυρία Πρόεδρε, κάποια πράγματα για τις σημαντικές προόδους που έγιναν ε, στον νομοθετικό τομέα. Πρόσφατα ε, ψηφίστηκε ο νόμος 1309 ε, που αυξάνει την ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία ε, μέλους συνδικαλιστικού, ε, συνδικαλιστικής ε, οργάνωσης από 20 σε 30 χρόνια. Και οποιαδήποτε παρεμπόδιση τη ελευθερίας του συνεταιρίζεσθε επιφέρει ποινικέ κυρώσεις. Συνεπώς λοιπόν δεσμευόμαστε στην οδό της βελτίωσης ε, η βελτίωση του Προέδρου ήταν ξεκάθαρες. Πρέπει να μειώσουμε το δίκτυο αυτό στο μηδέν. Θα πρέπει να μειώσουμε επιτέλους τη βία στην Κολομβία και για να το πράξουμε εφαρμόσαμε την πολιτική δημοκρατική ασφάλεια στη χώρα. Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι οι εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είναι αρκετά ξεκάθαρες, γιατί επισημαίνουν ακριβώς τις προόδους που σημείωσε η Κολομβία όσον αφορά την προστασία των συνδικαλιστών. Η χώρα είναι ανοιχτή στις ε, επισκέψεις μελών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, μέλη της Διεθνούς Συνομοσπονδίας ε, ε, συνδικάτων ή οποιαδήποτε άλλης, οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης που επιθυμεί να έχει κάποια στοιχεία ή πληροφορίες από εμά. Και ζητούμε από την άλλη πλευρά και δική σας υποστήριξη και δική συνεργασία για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενωμένοι, ούτως ώστε να μειώσουμε αυτά τα φρικιαστικά νούμερα. Ε, σας καλούμε λοιπόν σε διαβούλευση με την κυβέρνηση και τις ε, ε συνομοσπονδίες των εργαζομένων. Θα ήθελα να σας πω πως λοιπόν, στις 17 Σεπτεμβρίου ε, συνήλθαν ε, οι ενώσεις ε, συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζόμενων και προέβησαν σε μια κοινή δήλωση η οποία αποτελεί από 8 σημεία. Στο πέμπτο σημείο απορρίπτει κάθε μορφή, καταδικάζει κάθε μορφή βίας. τον Ιανουάριο αυτού του έτους υπήρξε, συντάχθηκε ένας ε, κοινός, ένα κοινό κείμενο μεταξύ κυβέρνησης και ενώσεων εργαζομένων για να υπάρξει κοινό μέτωπο κατά της ε, βίας την οποία ε, βιώνει η χώρα μας. Ε, επαναλαμβάνω, ήταν η Συνομοσπονδία Εργαζομένων της Κολομβίας ο χρόνος σας έχει τελειώσει, λέει η Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα λοιπόν, λέει ο μιλητής, να σας ε, ευχαριστήσω για την ε, ευκαιρία που μας δώσατε και να σας πω ότι ελπίζω στη διεθνή συνεργασία ούτως ώστε να παλέψουμε από κοινού κατά της μάστιγας αυτής που πλήττει την Κολομβία. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις των βουλευτών. Το λόγο έχει ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή τη σημαντική συνάντηση για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Κολομβία που θεωρώ ότι, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο. Ο, η Κολομβία είναι ένας θεματικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του πολιτικού διαλόγου και εφαρμόζεται το, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα. Εγώ ίδιο είχα το προνόμιο να είμαι επικεφαλής της, παρατήρησης, της ομάδας αντιπροσωπής παρατήρησης των εκλογών κάτω από πολύ δυσχερείς ε, συνθήκες και είχα την ευκαιρία να συζητήσω με το Μαρουλάνκα ε, και την στατική ομάδα του Φάρκα. Επίσης, υπέγραψα το ψήφισμα αυτού του Κοινοβουλίου που ζήτησε από το Συμβούλιο Υπουργών να συμπεριληφθεί το ΦΑΡΚ στον κατάλογο τρομοκρατικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο μας, κυρία Πρόεδρε, χρειάζεται να το επαναλάβω, έχει δεσμευθεί απολύτως για την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Κολομβία και παντού αλλού. Είναι προφανέ ότι τα στοιχεία που κατατέθηκαν εδώ δείχνουν μια σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να σα επενθυμίσω ότι η Σύνοδο των Επικεφαλήν Κυβερνήσεων στη Βιέννη δίνει μια εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρουσιάσει ορισμένε οδηγίε διαπραγματεύσει, ούτω ώστε να γίνει μια συμφωνία ε, ελεύθερου εμπορίου με την ε, ε, Κολομβία. Επίσης θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι αυτό το Κοινοβούλιο ενέκρινε τέσσερα ψηφίσματα και ε, ούτε ώστε να περατωθούν οι εμπορικές αυτές ε, συμφωνίες κατά την προσεχή σύνοδο της Μαδρίτης. Νομίζω ότι οι αριθμοί ε, μας δείχνουν ξεκάθαρα τα πράγματα. Είπαμε ότι υπάρχει μια απόκληση όσον αφορά τον αριθμό των 28 ή 40 συνδικαλιστών που δολοφονήθηκαν. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ακόμα και ένας συνδικαλιστής να δολοφονηθεί, αυτό είναι κάτι συνιστά μια απαράδεκτη πράξη. Ο εκπρόσωπος του συνδικάτου νομίζω εξέφρασε τα πράγματα πολύ σαφώς είπε ότι αυτή η κατάσταση που υπάρχει στη χώρα θα πρέπει να μας οδηγήσει στην ε, ολοκλήρωση της ε, εμπορικής συμφωνίας. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν άδικο εξετάζοντας τις προσπάθειες της ε, Κολομβίας όσον αφορά την πάλη κατά της τρομοκρατίας και την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το καταδεικνύει σαφώς η ειδική συγγήτρια για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία το Σεπτέμβριο αυτού του έτους νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικά άδικο να, να τιμωρήσουμε την Κολομβία για μια κατάσταση στην οποία είναι θύμα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των συνδικαλιστών στην Κολομβία. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει κυρία Πρόεδρε, πώ θα πρέπει να συμβάλλουμε ε, στο πλαίσιο αυτού του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να ολοκληρώσω, γιατί μα είπατε να είμαστε σύντομοι, ε, θέτοντα μία ερώτηση στον κ. Βανέρα. Κατάλαβα ότι η εργατική ότι 18 εκατομμύρια εργαζόμενων είναι στον ιδιωτικό τομέα και μόνο ένα εκατομμύριο των εργαζομένων εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν όλοι οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων συμμερίζονται τη δική σας άποψη, γιατί θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη των εκπροσώπων, των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα περιοριστούν οι επόμενες παρεμβάσεις στα δύο λεπτά. Τον λόγο έχει ο κύριος Μέντε Δεβάγε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμμερίζομαι το σύνολο των ε, επιχειρημάτων του κυρίου Σαλαφράγκα και θα ήθελα να σας πω το εξή, όσο, όσο μεγαλύτερη ακριβία γίνεται. Καταρχήν, η κυβέρνηση της ε, Κολομβίας, ή μάλλον καλύτερα, το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να σα παρουσιάσω εδώ είναι το εξή. Η κατάσταση είναι δυσχερή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία και ιδιαίτερω ευαίσθητη. Ωστόσο υπήρξε χειρότερη ε, και πιο ευαίσθητη στο παρελθόν. Ε, είναι προφανές ότι υπάρχει μια θετική διαδικασία προς τα μπρος. Δεύτερον, η κυβέρνηση της Κολομβίας αναγνώρισε τα σφάλματα ε, που σχετίζονται με αυτή την κατάσταση. Υπήρχαν περισσότερα σφάλματα στο παρελθόν από ό,τι στο παρόν τα αναγνώρισα σφάλματα. Η κυβέρνηση Κολομβίας είχε τη δυνατότητα να κάνει μια έκκληση μάλλον έχει γίνει μια έκκληση, συγγνώμη, προ την κυβέρνηση τη Κολομβία, ούτω ώστε να προσπαθήσει να αυξήσει την αξιοπιστία τη. Και ο μόνο τρόπο να αυξηθεί η αξιοπιστία τη κυβέρνηση είναι να ε, πάρει συγκεκριμένα μέτρα κατά τη βία. Θα ήθελα να σας να αναφερθώ σε τρεις ε, προκλήσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό η κυβέρνηση της Κολομβίας να αντιμετωπίσει το, ε, θέμα των περιπτώσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Νομίζω ότι θα πρέπει να προθεθεί ο νόμος για τα θύματα της ε, τρομοκρατίας, νόμος ο οποίος ε, τελικά, ενώ πρόκειτο να εγκριθεί, τελικά απορρίφθηκε, γιατί θεωρήθηκε ότι είχε υψηλό πολιτικό κόστος. Και Τρίτον, είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση της ε, Κολομβίας να προχάγει ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε συνένεση με την κοινωνία των πολιτών. Εάν αυτό γίνει από την κυβέρνηση της Κολομβίας θεωρώ ότι θα αποτελέσει μια θετική χειρονομία και θα οδηγήσει περισσότερους ε, ευρωβουλευτές να τεθούν υπέρ της σύναψης εμπορικής συμφωνίας με την Κολομβία. Γιατί η συμφωνία αυτή θα δεσμεύσει την κυβέρνηση ούτως ώστε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Κάσμαν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Όντως έχουν γίνει κάποιες πρόοδοι, αλλά έχω και σημαντικές ανησυχίες βέβαια. Το να λέμε τώρα ότι έχουν μειωθεί οι θάνατοι και ότι έχουν περάσει, έχουμε φτάσει στους 40, μα ναι, είναι 40 όμως δολοφονίες που θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Εγώ και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου στο εργατικό κόμμα της Τμήματου ε, Βασιλείου πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να εγκριθεί μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω διάλογος πρέπει να γίνουν περισσότερες συζητήσεις. Το επιχείρημα είναι ότι χωρίς την συμφωνία αυτή ή μάλλον με τη συμφωνία αυτή θα βελτιωθεί η ζωή των συνδικαλιστών δεν έχουμε τη συμφωνία και από την άλλη η κυβέρνηση μας λέει ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση των δικαλιστών. Εγώ θεωρώ ότι περιμένοντας να υπογραφεί η συμφωνία αυτή ή μάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή προκειμένου να γίνουν περισσότερες αλλαγές, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται από την κυβέρνηση και από τον νόμο. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στην εφαρμογή των αρχών μας, ιδίω όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαφορετικά βάλουμε κατά τον ίδιο των αρχών μας. Είτε οι αρχέ αυτέ εντοπίζονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εκτό. Και, κυρία, ε, και τέλο, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω και είμαι στη διάθεσή σα για να πείτε το αντίθετο ότι ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε ο Καναδά, ούτε η Νορβηγία δεν έχουν επικυρώσει τη συμφωνία του. Φαίνεται ξαφνικά ότι θα σπάσουμε την αλληλεγγύη μα με άλλου σημαντικού εμπορικού μα εταίρου, ενώ θα μπορούσαμε να εργαζούμε μαζί του προκειμένου να πετύχουμε καλύτερε αλλαγέ και προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Κολομβία. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βάλουμε κατά τη λυγή που έχουμε με τι άλλε χώρε. Στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θέλω φίλου, θέλω αλλαγέ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μίτσελ για την οργάνωση αυτή τη συνάντηση. Να σας υπενθυμίσω κάποια συμβάντα στα οποία αναφερθήκαμε. Το 2009 ανανεώθηκε η απονομή, αν θέλετε, στην Κολομβία μετά την υπογραφή 27 συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον της ιδιότητας των, του καθεστώτος των γενικευμένων προτιμήσεων. Το 70% των συνδικαλιστών στον κόσμο που φωνεύονται, φωνεύονται στην Κολομβία, μπορούμε δυστυχώς να μιλήσουμε για γενοκτονία πολιτική. Βέβαια χρόνο με τον χρόνο ε, μειώνονται λιγότεροι συνδικαλιστές, απλούστατα γιατί μειώνεται γενικά ο αριθμός τους, στο τέλος δεν θα μείνει κανείς οι Αμερικανοί Δημοκράτες ήδη από το 2006 έχουν μπλοκάρει κάθε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Κολομβία και είπαν ότι για να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία ε, απαιτείται ασφάλεια για τους εργαζομένους και προστασία του περιβάλλοντος. Μπροστά σε αυτές τις μορφές των παραβιάσεων στη Σρι Λάνκα, το καθεστώς της ετορικής σχέσης αφαιρέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Σρι Λάνκα. Και τελευταίο συμβάν το οποίο πρέπει να υπογραμμίσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά μια τράπεζα τεχνικών διαπραγματεύσεων με την Κολομβία και το Περού. Δύο χώρες οι οποίες στη Λατινική Αμερική σέβονται λιγότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατανοούμε βέβαια την επιθυμία της Ισπανικής Προεδρίας να παρουσιάσει υπογεγραμμένες συμφωνίες στις 17 και 18 Μαΐου στη Μαδρίτη αλλά θα ήθελα να ζητήσω επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει έρευνα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία όπως το έκανε στη Σρι και να διακόψει τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία αν δεν υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι ντροπή για μας που υποτίθεται έχουμε την φιλοδοξία να προασπιζόμεθα τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αγνοούμε το πρόβλημα και να κάνουμε λιγότερο από ό,τι οι συνάδελφοί μας τη ΣΥΠΑ. Κύριος Χάουιτ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γκέι Μίτσελ. Ελπίζω να υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για άλλες χώρες τέτοιου είδους συζητήσεις δηλαδή. Εγώ συνδέομαι με την εκστρατεία για τη δικαιοσία στην Κολομβία όχι μόνο για τους συνδικαλιστές αλλά για όσους προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λέγουν ότι τα δύο τρίτα των θανάτων που προκαλούνται από τα συστήματα ασφαλείας των χωρών σημειώνονται στην Κολομβία. Ο Υπουργός μας είπε ότι θέλει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και να μειωθεί ο θάνατος, να μειωθούν οι θάνατοι των συνδικαλιστών. Πώς μπορείτε από τη μία να υπογράψετε τα, τις συμβάσεις αυτές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρμόζετε τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται. Για, το διεθνές, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας πράγματι σας ευχαριστούμε για τα παραδείγματα που δώσατε. Είναι λίγα τα παραδείγματα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να καλύψει ε, τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στην νομοθεσία από τη μία και την εφαρμογή της από την άλλη. Είπατε ότι παίρνει νέα μέτρα η κολομβιανή κυβέρνηση για να αποτραπούν τρομοκρατικές ενέργειες και πράξεις βίας εις βάρος των συνδικαλιστών και των εκπροσώπων των εργαζομένων γενικότερα. Πιστεύετε εσείς ότι το κράτος που είναι εν μέρη υπεύθυνο για τις δηλοφονίες μπορεί να πάρει αυτά τα μέτρα και είναι αλήθεια το ότι τα δύο τρίτα των θανάτων των συνδικαλιστών ε, εμπλέκονται στα δύο τρίτα και δομές του Κολομβιανού κράτους. Δύο επιπλέον σημεία. Γιατί όπως μας είπε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας χρηματοδοτήσατε προγράμματα, δεν χρηματοδοτήσατε μάλλον προγράμματα που να έχουν του συγκεκριμένο στόχο το θέμα που συζητάμε σήμερα και τι σας εμποδίζει να το κάνετε αυτό στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών στο μέλλον. Για τον κύριο Κάσμαν, γιατί δικαιολογείται το να συνεχίσουμε ε, την πορεία προς τη συμφωνία αυτή όταν η ΙΠΑ, ο Καναδάς και άλλες χώρες δεν το κάνουν αυτό για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν αξίζουν ενώ σε άλλες ναι. Ο Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι εγώ εκτιμώ και πιστεύω στις προσπάθειες που μας περιέγραψε ο Υπουργός της Κυβέρνησης όσον αφορά την πάλη κατά της ε, βίας τον αγώνα κατά της βίας. Το πιστεύω, αλλά οι αριθμοί δεν μας αφήνουν ε, πολλές ε, ελπίδες ε, ή πολλά περιθώρια ελπίδες. Μιλάμε για το 60 των δολοφονιών των συνδικαλιστών σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι δραματική ε, είναι κάπως βελτιωμένη, αλλά παραμένει αποτρόπαιη, αποκρουστική. Ε, Βεβαίω, μα είπατε ότι οι συνδικαλιστέ είναι μια κατηγορία. Είναι σαφέ ότι αποτελούν μια κατηγορία μεταξύ άλλων κατηγοριών που πάσχουν, υπέφτουν θύματα αυτή τη βία. Ε, εν πάση περιπτώσει, όπω είπα, εμπιστεύομαι τι καλέ προθέσει των αρχών της Κολομβίας. Παρ' αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να πετύσουμε πολύ περισσότερα και πιο ορατά ή πιο συγκεκριμένα καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ ήμουν φίλος του Χωσέ Μερκάδο, που ίσως θα τον γνωρίζετε. Ήταν ένας από τα βασικά ηγετικά στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος. Ε, δεν είχε δημόσιο αξίωμα, ήταν επικεφαλής του Συνδικάτου των Μουσικών στην Κολομβία και έπεσε επίσης θύμα του της ε, τρομοκρατίας ε, αφού είχε εκπροσωπήσει την ε, χώρα του και τα συνδικάτα πολλά χρόνια στη συνεδρία της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Είναι, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καινούριο φαινόμενο εδώ. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαρκεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Εγώ όπως σας είπα εκτιμώ να γνωρίζω τη βούληση να πατάξετε αυτό το φαινόμενο. Αλλά θα πρέπει να απαιτήσουμε να γίνουν περισσότερα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας ε, στην οποία αναφερθήκαμε και νομίζω ότι αυτό είναι συνεπές με τα όσα σκέφτομαι. Και ε, όταν μιλάμε για άλλες χώρες, για την Αμερική, εκεί οι νεκροί ε, δεν είναι χιλιάδες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τις αρχές αυτές της χώρας στην προσπάθειά τους. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο με σοκάρει εδώ με σοκάρει όταν μιλούμε για τις Ηνωμένε Πολιτείε ως ε, μοντέλο για μας, ως υπόδειγμα, επειδή αναστέλουν την ε, Συμφωνία Ελεύθερων ε, Συναλλαγών με την Κολομβία. Θα ήθελα να μας εξηγήσει ο κύριος Υπουργός πώς ε, η χώρα η οποία είναι ο βασικός ε, εταίρος του στον κόσμο δεν επικυρώνει αυτή τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Δέχομαι, όπως είπα στην αρχή, ότι έχουν υπάρξει βήματα προόδου. Αναγνωρίζω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κολομβιανή κυβέρνηση. Προέρχομαι από ένα νησί όπου για 30 χρόνια ο κόσμος σκοτωνόταν και κατανοώ το πρόβλημα του ελέγχου της τρομοκρατίας, αλλά βλέπουμε εδώ. Από τους 250 το 91 μέχρι τους 37 το 2009 είναι φυσικά βήματα πρόοδου. Βέβαια δεν ξέρω τι έγιναν το 2004 με το 2007-2008 γιατί είναι σαφές ότι και εκείνα τα χρόνια δολοφονήθηκαν οι ηγέτες των συνδικαλιστών. Γιατί έγινε αυτό, γιατί διεκδικούσαν καλύτερες αξιοπεπέστερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβέ και αυτό είναι απαράδεκτο. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και προς την κυβέρνηση και προς τον Υπουργό και όποιον εμπλέκεται γενικότερα με τα θέματα αυτά. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Και ο λόγος για τον οποίο συζητάμε τα θέματα αυτά σήμερα είναι γιατί θεωρούμε γενικά τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι θα γινόταν είχαν σκοτωθεί ας πούμε 23 συνδικαλιστές στην Νορβηγία, τη Γαλλία ή τη Γερμανία το 2009. Λοιπόν, αναγνωρίζουμε ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά το πρόβλημα παραμένει πάρα πολύ σημαντικό. Τα στοιχεία που μας μετέφερε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η σχέση ανάμεσα στον διάλογο αυτό και την άμεση αναπτυξιακή βοήθεια ε, Έχουμε μια ομάδα η οποία ασχολείται με το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας προς τις χώρες της περιοχής και θα τους ενδιέφερε να ακούσουν τι στοιχεία έχετε. Μας έχετε διανύμει και απευθύνομαι στον πρέσβη ή τον Υπουργό σχετικά την έκθεση του Αμερικανού αντιπροσώπου όταν επισκέφθηκε την Κολομβία. Και τίθεται εδώ το θέμα της προστασίας των συνδικαλιστών ηγετών από σωματοφύλακες, τους οποίους θα πληρώνει η κυβέρνηση. Οι τρομοκράτες ε, δολοφονούνται, ε, δολοφονούν μάλλον άκρητα και δεν νομίζω ότι μια τέτοια μορφή προστασίας θα ήταν η λύση για το πρόβλημα. Εδώ κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών γιατί δεν έχουμε πλέον χρόνο στη διάθεσή μας, λέει η κυρία Ζολή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Μίση, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ προσυπογράφω τα όσα είπε ο κύριος Σαλαφράνκα και την ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυρίου Μαρτίνεθ. Αυτή η συμφωνία ε, δεν είναι ότι η Ισπανία θέλει να πετύχει κάτι εντός της ε, προεδρίας της. Ε, το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθεί μια διαδικασία την οποία διαπραγματευόμαστε εδώ και τρία χρόνια βάσει μιας εντολής που μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ώστε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία που εμεί ήδη ξεκινήσαμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Κολομβία υποβάλλεται σε μια σειρά ελέγχων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διεθνέ επίπεδο. Το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ασκεί αυτού του ελέγχου και η συμπεριφορά τη όσον αφορά την προσπάθεια ε, πάταξη της ε, βίας είναι σύμφωνη με μια σειρά διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Κολομβία και η οποία προσπαθεί να τι εκπληρώσει σε κάτω από δυσχερεί συνθήκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει τι ε, συμφωνίε με το Ουσμπεκιστάν και την ε, Γεωργία και προσπαθούμε να ανοίξουμε κάποια κανάλια με τον τρόπο αυτό διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας σε ολόκληρο τον κόσμο, εντό του πλαισίου της διεθνούς κοινότητας. Εάν δεν έχουμε καμία συμφωνία με την Κολομβία, είναι πολύ δύσκολο να ασκήσουμε μια επιρροή όσον αφορά τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τρομοκρατούν οι στατιστικές αυτές, τα στατιστικά δεδομένα που ακούσαμε για δολοφονίες και άλλες εγκληματικές πράξεις. Είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης αυτοί οι οποίοι αναφέρονται στα στατιστικά αυτά δεδομένα και προσπαθούν να εξηγήσουν τη διαφορά από, τη μια, από, την, από τον αχρόνο στον άλλον. Επομένως, η κυβέρνηση είναι αυτή που θα πρέπει να μας ε, πει τι περιμένουν από τις δικέ του αρχέ, ποια είναι τα δικά του στατιστικά δεδομένα, δηλαδή τι έχει κάνει η αστυνομία, τι έχουν κάνει οι δικαστέ, πόσους τελικά έχουν συλλάβει, πόσου έχουν καταδικάσει, γιατί Το κράτος δικαίου υφίσταται μόνο αν είμαστε σε θέση σε μία χώρα να εμπιστευτούμε τις αρχές εκείνες επιβολής της τάξης που βάλλονται κατά της εγκληματικότητας. Έρχομαι από την ε, περιοχή των Βαλκανίων και χωρίς τα δικαστήρια, χωρίς ένα δικαστικό σύστημα, αν δεν είχαμε καταφέρει να συλλάβουμε και να τα καδικάσουμε υπεύθυνου, το μόνο που θα είχαμε στα χέρια μας θα ήταν στατιστικά δεδομένα για τους θανάτους, για τα θύματα, για τις δολοφονίες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι καταδικάζονται άνθρωποι για τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει, ότι οι προδιαγραφές, αν θέλετε, για την καταπολέμηση του εγκλήματος έχουν ε, αυξηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι τα στατιστικά δεδομένα των αρχών επιβολής ε, του νόμου. Ο κύριος Φίλς Εξελά, ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές που παρουσίασαν αυτά τα στοιχεία. Μου άρεσε που είχαμε την ευκαιρία επίσης να ακούσουμε τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους που παρίστανται εδώ, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε και τους, υπαλλήλους, ε, τους υπολείπους συγγνώμη, που δεν, έπερα, ε, δεν πήραν το λόγο. Όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως μας είπε ο κ. Υπουργό, είναι δυσχερής. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε τις σημαντικές βελτιώσεις που σημειώθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση. Από αυτέ τις 40 ας πούμε δολοφονίε των συνδικαλιστών, πόσοι από του συνδικαλιστέ δολοφονήθηκαν για την συνδικαλιστική του δραστηριότητα. Νομίζω ότι είναι μόνο μία τέτοια περίπτωση και όπως φαίνεται το άτομο αυτό δολοφονήθηκε από το ΦΑΡΚ, όπως είπαν οι δικαστικές αρχές. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια σύγκριση με άλλες ε, χώρες. Εγώ είμαι καινούριο σε αυτό το σώμα, αλλά θα ήθελα να σε επενθυμίσω ότι στην προηγούμενη θητεία υπογράφηκε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Μεξικό, με την κυβέρνηση Βιλπρί, που είναι αριστερή. Και εγώ δεν θα ήθελα να εφαρμόσουμε εδώ την αρχή δύο μέτρα και σταθμά. Δηλαδή, να έχουμε μια συγκεκριμένη στάση με μια κυβέρνηση μόνο και μόνο επειδή είναι αριστερή και μια διαφορετική με μια κυβέρνηση που δεν είναι αριστερή. Θα ήθελα να σας πω αυτό που είπε ο Αλμπέρτο Μπουνόρη το Μοξικό, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναλύσαμε διάφορα μοντέλα και πιστεύουμε ότι το μοντέλο της Κολομβίας είναι το πιο ενδεδειγμένο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ας μας χρησιμεύσει σαν ένα δείκτης για τις σημαντικές βελτιώσεις που σημειώθηκαν στην Κολομβία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνο ε, θα πάρει το λόγο για τη Λατινική Αμερική της Διεύθυνσης Ρελέξ για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ανησυχητική η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυβέρνηση του Ρίμπε έχει κάνει προσπάθειες για την επικράτηση του κράτους δικαίου και εν μέρη οι προσπάθειες αυτές ήσαν επιτυχείς. Όμως οι φόνοι και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τις ε, τα δίκτυα διαλόγου τα οποία έχει για να προσπαθήσει να προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα αυτούς που προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους συνδικαλιστές. Προσπαθούμε επίσης να στηρίξουμε τις προσπάθειες μείωσης της ασυλίας ή ατιμορρησίας, η οποία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Δείχνουν οι τελευταίες έκθεσεις, εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών ότι πολλά μένει να γίνουν και η κυβέρνηση έχει κάνει κάποιες αλλαγές στο νομικό σύστημα στοιχειοθετούνται θετικές λοιπόν εξελίξεις στον τομέα της δυνατότητας δημιουργίας νέων συνδικάτων και οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν. Εμείς θα πάρουμε μέρος στην προσπάθεια συντονισμού της βοήθειάς μας προς την κατεύθυνση αυτή. Προωθήσουμε γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων επίσης στην Κολομβία. Ε, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Κολομβίας μέσω του πολιτικού διαλόγου, μέσω του διαλόγου του συγκεκριμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του προγράμματος οικονομικής συνεργασίας. Είμαστε σε επαφή επίσης και με την Σκουέλα Nacional Συνδικάλ, μια πολύ σεβαστή παγκοσμίως συνδικαλιστική μη κυβερνητική οργάνωση. τα 30 εκατομμύρια από τα 160 τα οποία θα δοθούν στη χώρα αυτή στην περίοδο 07-013 έχουν σαν στόχο την επικράτηση του κράτους δικαίου. Ταυτόχρονα η Κολομβία χρειάζεται την οικονομική ανάπτυξη για να μειωθεί η απασχόληση, να μειωθεί ο γκρίζος τομέας της οικονομίας θεωρούμε ότι η πολυμερής εμπορική συμφωνία την οποία διαπραγματευόμεθα με τη Δημοκρατία της Κολομβίας έχει την δυνατότητα να συνεισφέρει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε η συμφωνία να περιλαμβάνει μία ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρέποντας και την μονομερή διακοπή ισχύω της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα Θέλουμε να περιλαμβάνονται ορισμένε δεσμευτικές αναλήψεις υποχρέωσης σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προτείνουμε και έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογή του εργατικού δικαίου μέσω των οργανώσεων και των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών. Όλα αυτά είναι ένα νέο θετικό βήμα για την προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης στην Κολομβία και της τύχης των συνδικαλιστών ιδιαίτερα. Οι ομιλητές λοιπόν θα πρέπει να δώσουν σύντομες απαντήσεις, ένα λεπτό ο καθένας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Βανέγας. Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση αυτή σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των συνδικαλιστών. Oh, um, Είναι εκτός μικροφώνου η παρέμβαση. Ε, η πρόεδρος λέει επειδή ε, δεν έχουμε ε, κατεξαίρεση, επειδή δεν σας δώσαμε το λόγο, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν ζήτησα το λόγο επί τη ουσία γιατί αυτό το έπρεξαν οι συνάδελφοι Μαρία Μονίθ και Μίλιο Μενέντε. Ε, θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο προέχει σε αυτό το θέμα δεν είναι το υπόβαθρο αυτής της ε, προβληματικής, γιατί αυτό είναι προφανές. Νομίζω ότι ο κύριος Βανέκα γνωρίζει ότι αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται σε καμία άλλη τρίτη χώρα του κόσμου οι υπουργοί, οι συνδικαλιστές, οι πρέσβεις έχουν έρθει κατά επανάληψη εδώ και έχουν εξηγήσει την κατάσταση. Η Επιτροπή του Ερθρού Σταυρού κλπ. Είναι μια χώρα η οποία έχει αναλυθεί όσο καμία άλλη. Ε, εγώ είμαι σοσιαλιστής η κυβέρνηση της ε, Κολομβίας ε, είναι άλλη ιδεολογία. δεν έχω καμία απολύτω συμπάθεια για την κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζω ότι υποβάλλεται στον έλεγχό μας και στα δικά μας κριτήρια όσο καμία άλλη χώρα του τρίτου κόσμου. Ευχαριστώ. Κύριε Βάνεγκας, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Το πρώτο που θα ήθελα ήταν να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που έγινε αυτή η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ζήτημα της σύναψης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Κολομβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητιέται εδώ και τρία χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, εισακούμε τις ανησυχίες ε, που είναι σε διεθνές επίπεδο για τις δολοφονίες των συνδικαλιστών. Νομίζω είναι θέμα το οποίο δεν μπορούμε να επεκφύγουμε. Και θα ήθελα να σας πω ότι στην ε, Κολομβία θεωρούμε ότι πρόκειται για μια αληθινή τραγωδία. Προσπαθούμε να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστών. Υπήρξε μια απιστοχώρηση σε αυτές τις οργανώσεις, μια συρρήκνωση των συνδικάτων γιατί πριν από 15 χρόνια είχαμε 12% του ενεργού πληθυσμού που ήταν μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ τώρα ε, τα μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι μόνο 4% των εργαζομένων. Συνεπώς, λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα πλήγμα και κατά του συνδικαλισμού ε, εν γέννη. Ο στιγματισμός του συνδικαλιστικού κινήματος είναι συνεχής. Γι' αυτό θα ήθελα να σας εκφράσω τη διασύνδεση με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Ε, το πώς συνδέονται αυτά τα θέματα είναι κοινή άποψη της ε, Συνομοσπονδίας Εργαζομένων στην Κολομβία και ε, της κυβέρνησης. Ε, οι συνδικαλιστές, ε, οι δημοσιογράφοι ε, πέφτουν θύματα αυτής της βίας. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα διάλογο με το... Συνεργαζόμαστε με το Κομμάντο Νασιονάλ όσον αφορά τον, τις ελάχιστες αποδοχές, τον καθορισμό των ελάχιστων αποδοχών ενώ γιατί η κυβέρνηση με εντελώς απαράδεκτο και αθέμητο τρόπο δεν δέχεται αυτό το διάλογο εν σχέση και απορρίπτει την, τον καθορισμό του ελάχιστου μισθού των ελάχιστων αποδοχών. η κυβέρνηση μας έχει παρακάμψει απολύτως όσον αφορά το ζήτημα αυτό των ελάχιστων αποδοχών. Το λόγο έχει κυρία Ντούμπια Ονδρή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω σε τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη είχε να κάνει με τη δήλωση που έκανα για το αν ή όχι το κράτος της Κολομβίας ε, έδειξε υπεύθυνη στάση όσον αφορά την προστασία των ε, συνδικαλιστών. Κοιτάξτε, ένα κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει το δικαίωμα στην ζωή, σίγουρα, και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Κολομβία, η κυβέρνηση συζητούσε το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών προστασίας για τους συνδικαλιστές και για την επόσυρση των υπηρεσιών αυτών δεσμεύτηκε τελικά για την επέκταση και τη διατήρηση των υπηρεσιών αυτών προστασίας και εγγυήθηκε ότι ανεξάρτητα του τρόπου που θα χρησιμοποιούσε για την προστασία των συνδικαλιστών η κυβέρνηση ως κράτος, ως κυβέρνηση θα διατηρούσε την ευθύνη για την προστασία των συνδικαλιστών. Νομίζω ότι αυτό απαντά την ερώτησή σας. Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με το τι κάνει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας για το ζήτημα της ατιμορρησίας και τις σχετικές έρευνες. Κοιτάξτε, το ζήτημα της ατιμορρησίας αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα. Η υπόθεση 1787 που εξετάζει η Επιτροπή για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεστε του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και ζητήθηκε από την κυβέρνηση να ζήνουν οι απαραίτητες έρευνες από έναν εξάρτητο όργανο από μια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό άλλωστε απαιτείται από κάθε κυβέρνηση, κάθε φορά που υπάρχουν δολοφονίες, κάθε φορά που υπάρχει ατιμορρησία, οι έρευνες θα πρέπει να είναι σαφώς ανεξάρτητες. Και η κυβέρνηση της ε, Κολομβίας μέσω της ε, εισαγγελίας πρόκειται να διεξάγει την έρευνα αυτή με τρόπο ανεξάρτητο και οι ε, έρευνες αυτές, είπαμε εμείς στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ότι θα πρέπει να βελτιωθούν, θα πρέπει να ενισχυθούν και ότι θα πρέπει να εξεταστεί κάθε πτυχή των φαινομένων ατιμορρησίας που έχουν παρατηρηθεί στην Κολομβία. Ήρθαμε σε επαφή με την εισαγγελία και λάβαμε την πληροφορία από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν οι απαραίτητοι πόροι προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητε έρευνε στα πλαίσια τη υπόθεση 1787, προκειμένου στη συνέχεια το δικαστικό σύστημα στην χώρα να μπορέσει να προχωρήσει σε προσαγωγέ. Και τέλος, αναφέρθηκα στο ζήτημα της συνοχής που θα πρέπει να υπάρχει στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης. Όλοι οι οργανισμοί έχουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή να έχουμε μηδενική ανοχή όσον αφορά την παραβίαση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, μηδενική ενοχή όσον αφορά τις δολοφονίες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε με απόλυτη συνοχή και συνεκτικότητα, να φέρουμε μαζί τις δυνάμεις μας, τους πόρους μας, τις ικανότητές μας, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα βασικά ελλείμματα που ακόμα υπάρχουν στην ε, Κολομβία. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, αν υπάρχει η απαραίτητη οικοδόμηση εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση, τότε νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στο να προστατεύσουμε τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στην Κολομβία. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις της χώρας αυτής. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασία, αλλά και άλλοι οργανισμοί πιστεύω ότι θα πρέπει να συμβάλλουν. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σερικάντο Αντρέσε Σεβερή, Υπουργό Εργασίας, για δύο λεπτά. Ήθελα εξ ονόματο τη κυβέρνηση τη Κολομβία να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την κατάσταση στη χώρα μου και θα ήθελα εν συντομία να διατυπώσω ένα προβληματισμό τον εξή. Η πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι, είναι καθολική υπόθεση, οικουμενική υπόθεση. Τη συμμερίζεται η χώρα, η κυβέρνηση και η κοινωνία της Κολομβίας. Ε, στη χώρα μου είναι παρόντες όλοι οι πολυμερείς ε, οργανισμοί που έχουν προσκληθεί από την κυβέρνηση της Κολομβίας. Η, Κολομβία συνδέεται με όλα τα όργανα αυτά ε, τόσο από περιφερειακή όσο και από πολυμερή άποψη. Η Κολομβία είναι συνεχώς ανοιχτή στον διεθνή έλεγχο και στα σενάρια τα οποία έχει ορίσει η διεθνή κοινότητα. Για το λόγο αυτό η Κολομβία παρουσιάζεται με τη θέλησή της στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να υποβληθεί στον έλεγχο όλων των χωρών μελών των, της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό το λόγο η Κολομβία παρουσίασε μια έκθεση ε, παρακολούθησης των ε, δεσμεύσεων ε, τους προηγούμενους έξι, που αφορούν τους προηγούμενους έξι μήνες. υπάρχει ένας μηχανισμός διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του οποίου η ατζέντα είναι ουσιαστική και συμπεριλαμβάνει όλες τις ε, πτυχές των ανησιών που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνείδηση ότι η βελτίωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι ο καρπός ε, της ε, οριστικής ε, υπέρβασης της βίας που επηρεάζει όλους τους τομείς κοινωνίας της Κολομβίας εδώ και πολλά χρόνια. Υπό την έννοια αυτή κατανοούμε ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών που διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μηχανισμός κατά της βίας και κατά συνέπεια ένας δρόμος προς τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, για το λόγο αυτό, αφού επαναλάβουμε τις ευχαριστηρίες μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητούμε συνεργασία και μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους της Κολομβίας για την υπόθεση αυτή, την οποία σημεριζόμεθα. Ο Ξέρω ότι έχουμε τον Επίτροπο που έχει έρθει από την ΑΕΤ. Δεν θα ήθελα λοιπόν να αναλώσω πάρα πολύ χρόνο. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι κάναμε τη ζήτηση αυτή. Στόχος ήταν να επικεντρωθούμε στο σημαντικό αυτό ζήτημα και να εξασφαλίσουμε ότι η τάση αυτή που παρατηρείται για τη δολοφονία δηλαδή των συνδικαλιστών θα σταματήσει, θα σταματήσει εντελώς και θα αποτελέσει φαινόμενο του παρελθόντος. Αυτό περιμένουμε από όλα τα κράτη-μέλη και από όσες χώρες αποτελούν εμπορικούς εταίρους της Κολομβίας. Είναι σημαντικό ότι μιλήσαμε για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι θα πρέπει να επιτηρούμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή συστηματικά. Ναι, θα κάνουμε την επίβλεψη αυτή κύριε Μίτσελ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα με το υπόλοιπο της ημερήσιας διάταξης. Ένα δέκα δευτερόλεπτα παρακαλώ, μικρό διάλειμμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω δύο συμμετέχοντες στην εδρίασή μας που θα μας μιλήσουν για τον καταστροφικό σεισμό στην ΑΕΤ. Κύριε Μαρτίνες, παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, καθίστε. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω δύο συμμετέχοντες στη συνεδρίασή μας, όπου θα στήσουμε τον καταστροφικό σεισμό της ΑΕΤΙΣ, της 12ης Ιανουαρίου. Καταρχάς καλωσορίζω τον Επίτροπο Κάρελ Ντεγκούχτε και στη συνέχεια την Γκρέτα Σόμαντς, εκπρόσωπο της μη κυβερνητική οργάνωσης Συντονισμός Ευρώπη ΑΕΤ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε βέβαια το σημείο αυτό συζήτηση για την ΑΕΤ με μια πολύ λυπηρή είδηση για την οποία λάβαμε επιβεβαίωση όσον αφορά μια πρώην συνάδελφο του Κοινοβουλίου η οποία από το 2002 εργαζόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία όντας στην ΑΕΤ ήταν ε, το υπαριθμό 2 της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά αυτόν τον τρόπο συμμετείχε σε μία συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών στο Πόρτον Πραντς, όταν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνέβη ο σεισμός στις 12 Ιανουαρίου. Πρωτού συνεχίσουμε λοιπόν τη σύντηση για την Αιτή, θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν της συναδέλφου μας, η οποία εργαζόταν ακατάπαυστα για την ανθρωπιστική βοήθεια και η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας της, όπως τόσοι πολλοί κάτοικοι της ΑΕΤ, οι οποίοι πλήγησαν από το καταστροφικό αυτό σεισμό. Οι σκέψεις μας συνοδεύουν την οικογένειά της, η οποία υποφέρει. Ας συνεχίσουμε τώρα την συζήτησή μας για την ΑΕΤ. Η εξέλιξη κατάστασης εκεί είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Επιτροπή μας εξαιτία των διαστάσεων που έχει πάρει η δραματική κατάσταση στην ΑΕΤ και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 250.000 τραυματισμένους, 1,5 ε, εκατομμύρια αστέγων και 75.000 νεκρών. 112.000 νεκροί, με συγχωρείτε. Κατά τη διάρκεια τη έκτακτη συνεδρία Συμβουλίου των Υπουργών στι 18 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να δώσει 122 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική υποστήριξη και βοήθεια εκτάκτου ανάγκη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να δώσει 300 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υπάρξει μια άμεση ανοικοδόμηση και μια νοικοδόμηση συνέχεια ε, μεσοπρόθεσμη και, βράχη, και μακροπρόθεσμη, συγχωρείτε. Καταλαβαίνετε όμω ότι ε, η βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει οργανωτικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην ΑΕΤ και προβλήματα συντονισμού. Καταλαβαίνετε ότι ε, ενδεχομένω η κρίση αυτή να δώσει νέα όθηση στι πρωτοβουλίε που έχουν ξεκινήσει προκειμένου να γίνεται καλύτερος συντονισμό στις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας και άμεσα αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης μπορεί να δοθεί και νέα όθηση στο άρθρο 214 της Συνθήκης της Λισαβόνας, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία, προκειμένου να προωθήσει το συντονισμό ανάμεσα σε όλες τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, προκειμένου να διατίθεται εγκαίρως ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες που το έχουν ανάγκη. Θα ακούσουμε τον Επίτροπο Ντεγκούχ, το οποίο ε, ήταν στην Αιτή την προηγούμενη εβδομάδα και θα μας πει ακριβώς πώς έχει η ανθρωπιστική κατάσταση εκεί. Κύριε Ντεγκούχ, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. <coughs> Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, μόλις επιστρέψαμε από την Αιτή, είχαμε πάει σε μια αποστολή με πολλούς στόχους, θα έλεγα, Πρώτον να παρουσιάσει, πρώτον να καταθέσουμε τα συλληπιτήριά μας προς τον λαό της Αιτής και επίσης προς την οικογένεια της χιλίας Πιλάρ Σουαρές στην οποία αναφερθήκατε, την οποία μνημονεύσατε. Δεύτερον, προσπαθούσαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση επιτόπου αυτή την εποχή, γιατί υπήρχαν κάποιες αντιφάσεις ανάμεσα στις ε, εκθέσεις και τα στοιχεία που μας έδιναν οι συνεργάτες μας επιτόπου και οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών και επίσης ανάμεσα σε αυτά τα οποία βλέπαμε στην τηλεόραση και στον τύπο. Και τρίτον να συνεννοηθούμε με τις αρχές της ΑΕΤΙΣ για το πώς θα προχωρήσουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τρία σημεία να αναφέρω καταρχάς. Πρώτον να σας πω πως έχει η κατάσταση. Υπάρχουν προβλήματα κατεπήγοντα, κατά δεύτερον που δεν είναι μόνο ανθρωπιστικού τύπου και τρίτον η προσπάθεια ανοικοδόμησης. Πρώτον, η κατάσταση σήμερα επιτόπου. Θα έλεγε κανείς ότι δεδομένης της ευρύτητας της καταστροφής η κατάσταση θεωρείται σχετικά ικανοποιητική υπήρξαν σωστικές επεμβάσεις οι οποίες ε, έσωσαν πάρα πολλές ζωές ακόμα και χθες. Υπήρξαν ε, μέσα στη διάθεση των σωστικών συνεργείων. Χάρη στην παρουσία της Μινουστάδε εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπήρχαν ε, εξοπλισμοί των Ηνωμένων Εθνών επιτόπου και χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανισμοί αυτοί και επίσης ε, συνοδεύτηκαν και από ειδικού εξοπλισμούς για την ανείχνευση των εντοπισμών επιζώντων και έτσι μπορέσαμε να σώσουμε πολλές ζωές. Δεύτερον, η κατάσταση σε ιατρικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές ε, ιατρικές ομάδες παρούσες. Έχουν δημιουργηθεί πολλά ε, νοσοκομεία εκστρατείας Κάποια νοσοκομεία επίσης συνεχίζουν να λειτουργούν, κάποια τμήματα νοσοκομείων από την, από την ίδια τη χώρα και έτσι όλοι που έχουν ανάγκη από βοήθεια, από φροντίδα μπορούν να έχουν τη φροντίδα αυτή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε λίγες μέρες και σε λίγες εβδομάδες η προσπάθεια θα έχει τευματιστεί ίσα ίσα μπαίνουμε ακριβώς τώρα στη φάση της λεγόμενης ε, χειρουργικής πολέμου, θεάτρου πολέμου, σαν παράδειγμα ακροτηριασμοί και αυτοί οι ακροτηριασμοί απαιτούν να υπάρξουν ε, εγχειρήσεις στο μέλλον τους επόμενους μήνες γιατί απλά μέχρι τώρα η φροντίδα δίδεται προς αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη. Και τρέφω σεβασμό προς όλους αυτούς που εργάζονται και εργάστηκαν μέχρι τώρα μέρα και νύχτα με μεγάλη ταχύτητα, με τρομερή αφοσίωση που δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε αισθήματα θαυμασμού απέναντί τους. Η κατάσταση σε επίπεδο νερού και τροφίμων τώρα. Διανέμεται το νερό στα στρατόπεδα, σε αυτά τα ανεπίσημα κέντρα συγκέντρωσης που υπάρχουν στο Πόρο Πρένς, Επίσης διανέμονται τροφές. Το γεγονός ότι η κατάσταση σε επίπεδο τροφίμων ήταν ήδη τεταμένη πριν από το σεισμό οδήγησε στο να υπάρχουν στόκ τροφών, τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών επιτόπου ήδη πριν το σεισμό επαναλαμβάνω και αυτά διανέμονται τώρα. Αυτό δεν είναι σοβαρό πρόβλημα γιατί το λιμάνι άρχισε να λειτουργεί εκ νέου χάρη σε ένα απλό το τμήμα το οποίο τέθηκε σε λειτουργία. Οι δρόμοι δεν έχουν πάθει ζημιές, οι δρόμοι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι καλοί δρόμοι γιατί ποτέ δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργούν θα μπορούσε κανείς ε, να φανταστεί ότι θα υπάρχουν ε, ρήγματα στους δρόμους, ε, τρύπες, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και οι δρόμοι χρησιμοποιούνται. Και λειτουργεί επίσης και το αεροδρόμιο του Ποροπράς, με μεγάλη θα έλεγα πυκνότητα πτήσεων αν και υπάρχει μόνο ένας διάδρομος από προσγείωσης. Ω προ αυτό δεν υπάρχουν μεσοπρόθεσμα ή βράχυπρόθεσμα σοβαρά προβλήματα. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι κατεπίγοντος χαρακτήρα είναι οι άστεγοι, οι οποίοι κοιμούνται στα πάρκα, στις πλατείες, οι οποίοι είναι απροστάτευτοι. Υπάρχουν ε, βέβαια πολλά τέτοια στρατόπεδα θέλετε συγκέντρωσης, ανεπίσημα όμως, ε, τους πηγαίνουμε τροφές, τους πηγαίνουμε νερό, αλλά δεν προστατεύονται από τίποτα. Ε, προστατεύονται από ότι τους περίσεψε πια, ότι διέσωσαν και δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι οξύ, γιατί η θερμοκρασία είναι καλή και το κλίμα είναι καλό, δεν βρέχει, υπάρχουν, η θερμοκρασία είναι 28-30 βαθμοί, δεν υπάρχει υγρασία και μπορεί κανείς να ζήσει στην Ήπεθρο. Αλλά μέσα σε έξι μήνες θα ξεκινήσει η περίοδος των βροχοπτώσεων και αν δεν λυθεί το πρόβλημα πριν από την έλευση της ε, περίοδου αυτής, η κατάσταση θα γίνει δραματική. θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ειδικά στρατόπεδα προστασίας εσωτερικά εκτοπισμένων για 250.000 άτομα. Είναι εφικτό, δύσκολο βέβαια. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή σε ληφθούν οι αποφάσεις για την ανέγευση ενός τέτοιου στρατοπέδου. Απαιτούνται κάποιες εβδομάδες ως τη στιγμή που θα λειτουργήσει, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα επαναλαμβάνω. Δεύτερον, η κατάσταση του κράτους. Έγιναν συζητήσεις αρκετά ενδιαφέρουσες και σε βάθος τα έλεγα με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβερνήσεώς τους. Όλοι αυτοί συνεδριάζουν σε ένα αστυνομικό σταθμό, διότι είναι το μόνο που στέκεται όρθιο από πλευρά των δημοσίων κτηρίων. Ένα αστυνομικό σταθμό μιας μικρομεσαίας πόλης. Προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Έτσι κι αλλιώς ήταν οι δομές του κράτους αρκετά εύθραυστες, αλλά στο Πόρο Πρανς οι περιοχές όπου υπήρχε το Προεδρικό Μέγαρο, τα Υπουργεία, είναι οι περιοχές οι οποίες χτυπήθηκαν πιο άσχημα. Πρόκειται για την περιοχή Καρφούρ, εκεί ήταν το επίκεντρο του σεισμού και είναι περίεργο να δει κανείς ότι κάποιες περιοχές έχουν καταστραφεί πλήρως και κάποιες άλλες περιοχές δεν έχουν φυγεί καθόλου. Είναι περίεργο να καταλάβει κανείς ε, τι έχει γίνει ανεξάρτητα από την ποιότητα της κατασκευής. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι αν είχαν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα στην κατασκευή δεν θα υπήρχαν οι καταστροφές αυτές. Θα μπορούσε. Από την άλλη όμως, κτίρια όπως το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή ήταν σε μία γραμμή σεισμική ε, έχει σχεδόν καταστραφεί. Δεν είμαι αρχιτέκτονας, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο το να πει κανεί ότι οι ζημίε οφείλονται στην κακή κατασκευή των κτηρίων. Οφείλεται ε, κυρίως ε, στο πού χτύπησε ο σεισμός. Εν πάση περιπτώσει εξαφανίστηκαν όλα τα υπουργεία, ε, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια γρήγορης αποκατάστασης του κρατικού μηχανισμού το οποίο λειτουργεί με περιορισμένη ταχύτητα. Όχι ότι θα λειτουργεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα λειτουργεί. Έτσι ώστε οι αιτινοί να μπορέσουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια ανοικοδόμησης και γι' αυτό προτείναμε στην κυβέρνηση της ΑΙΤΙΣ να τους βοηθήσουμε σε επίπεδο κτηρίων, να τους δώσουμε σε μια πρώτη φάση containers, που θα χρησιμοποιούνται σαν κατοικία ή σαν χώρος λειτουργίας, γραφείων κτλ. για να επανεκκινήσει τη λειτουργία του ο κρατικός μηχανισμός. Είναι απαραίτητο αυτό και είναι απαραίτητο για να παραμείνει και επιτόπου η Μινουστάδ. Η Μινουστάδ έχει ένα τμήμα στρατιωτικό και ένα τμήμα πολιτικό, μη ένοπλο. Για να μπορέσει λοιπόν να λειτουργήσει το κράτος το ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει η πολιτική ηγεσία της Μινωστά σε συνεργασία με τον πυρήνα του κράτους της ΑΕΤ να μπορέσουν να λειτουργήσουν για να ληφθούν αποφάσεις όποτε αυτό χρειάζεται, αποφάσεις σαν παράδειγμα για το πού θα υπάρξουν αυτά τα στρατόπεδα, τα τρέν που θα χτίσουμε εμείς, γιατί σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει μηχανισμός λήψης απόφασης. Τρίτον, για αυτή την κατεπίγουσα βοήθεια η οποία δεν είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα και σε συνεργασία με την Αιτινή κυβέρνηση τις επόμενες μέρες θα αποστείλουμε μια αναγνωριστική ομάδα που θα αποτελείται από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και των κρατών μελών ήρθαμε σε επαφή με τα κράτη-μέλη και υπήρξαν ορισμένα κράτη-μέλη που θα βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη αναγνώριση, θα έλεγα, της κατάστασης το ταχύτερο δυνατόν. Τρίτον, υπάρχει το θέμα της ανοικοδόμησης. Στο Μορεάλ γίνεται αυτές τις μέρες μια συνάντηση των χωρών φίλων της ΑΕΤ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα και ο Σκούσνερ μας εκπροσωπεί Μιλήσαμε στο τηλέφωνο πριν από μια μισή ώρα. Η βασική ιδέα είναι να υπάρξει ένα πραγματικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση της IT, των υποδομών της IT και του κράτους. Δεν πρέπει μόνο να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση των ζημιών του σεισμού, αλλά θα πρέπει να καλύψουμε αν θέλετε και ε, τα κενά τα προφανή τα οποία έχει ε, αυτή τη στιγμή το κράτος. Βασική ιδέα είναι λοιπόν να υπάρξει μια έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί στη συνάντηση των δωρητριών χωρών που θα γίνει σε δύο-τρεις μήνες, η λεγόμενη Pledging Conference. Είναι η συνάντηση ανάληψης υποχρεώσεων από πλευράς των δωρητριών χωρών, Pledging Conference και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η διάσκεψη αυτή και μάλιστα κάποιες χώρες που θα πάρουν μέρος όπως ο Καναδάς και η Δομινικανή Δημοκρατία που είναι γειτονική χώρα. Και η ΕΠΑ φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ορίσουμε το ταχύτερο δυνατόν κάποιον για να μας αντιπροσωπεύσει σε αυτή την προσπάθεια. Ένα ερώτημα, Πρόεδρε, σχετικά με την περιορισμένη εικόνα η οποία υπάρχει για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί, αλλά εκπροσωπείται μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών που εργάζονται εκεί δεν αναλαμβάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες δράσεις. Χρηματοδοτεί οργανώσεις οι οποίες εργάζονται για μας, με τα δικά μας χρήματα. Θα έλεγα ο στρατός δεν αποτελείται από υπαλλήλου της Επιτροπής και γίνονται επίσης προσπάθειες από όλα τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα από ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία έκαναν τεράστιες προσπάθειες και είναι παρούσες οι χώρες αυτές εθνικά θα έλεγα. Μια τρίτη παρατήρηση που εξηγεί την περιορισμένη σε εισαγωγικά ορατότητα βλέπουμε την αμερικανική ε, παρέμβαση σε επίπεδο στρατιωτικό. Πάρα πολύ. Βλέπουμε όμως ε, λιγότερο την ευρωπαϊκή παρέμβαση η οποία είναι σε επίπεδο ιατρικό, ανθρωπιστικό, χειρουργικό είναι πολύ σημαντική αν και λιγότερο εμφανής. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ντρέπεται κανείς σε εισαγωγικά για αυτά τα οποία κάνουμε στην περιοχή. Η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι πολύ σημαντική και υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα ορατότητας εντός εισαγωγικών, αλλά το θέμα το οποίο ανακύπτει είναι ακριβώς η ορατότητα αυτή ή η παρουσία επιτόπου. Νομίζω ότι εδώ δεν θα πρέπει να Εποταχθούμε στη λογική των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι ε, το πιο βασικό είναι τα θύματα και το πώς μπορούμε να τα συνδράμουμε στη δυστυχία τους. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενημέρωση των όσων γνωρίζουμε για την IT. Από εσά που έρχεστε από αυτή τη χώρα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σάλμανς για, δέκα 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης για την ε, πρόκληση στον συντονισμό ε, Ευρώπη-ΑΕΤ που είναι μια συνένωση πολλών μη κυβερνητικών οργανισμών που εργάζονται με 100 περίπου οργανώσεις, ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές οργανώσεις κλπ, οργανώσεις των αγροτών στην ΑΕΤ. Ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία μας συντονισμού το 2004 και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε την απήχηση που έχουν οι συστάσεις μας στην ΑΕΤ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις χώρες που παρίστανται εδώ για την μεγάλη αλληλεγγύη που επέδειξαν ε, μετά από αυτή την έκκληση βοήθειας για την ΑΕΤ και οι εταίροι μας εκεί είναι πολύ βαθύτερα συγκινημένοι από αυτή την αλληλεγγύη. Ωστόσο, η έκκλησή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες ε, μέλη έχει σαν στόχο να υπογραμμίσουμε ότι σε κάθε μορφή βοήθειας που παρέχεται και την ε, μορφή κατεπίγουσας βοήθειας επίσης ε, συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι δεν θα πρέπει να ε, παραμελούμε να συμπεριλαμβάνουμε την ε, κυβέρνηση ΑΕΤ και όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα διαφήματα και σε όλες τις πρωτοβουλίες ε, που γίνονται εκεί. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να διαγραμματίσουν ένα κεντρικό ρόλο όσον αφορά την ε, εκπόνηση των ενδεδειγμένων ε, δομών που θα επιτρέψουν την ανοικοδόμηση της χώρας και ιδιαίτερα του Πορτοπρένς και των ζωνών που έχουν πληγεί περισσότερο. Όσον αφορά την ε, βραχυπρόθεσμη απόκριση, νομίζω, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε το συντονισμό όλων των προσπαθειών υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών που συντονίζει την διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια. Και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να διαρματίσει εδώ ένα σημαντικό ρόλο για να επιμείνει ούτως ο συντονισμός αυτός να γίνεται πάντοτε σε σύνδεση με τους τοπικούς ε, οργανισμούς, τοπικές οργανώσεις και την κυβέρνηση της ΑΕΤ, έστω και αν είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένη αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι η άσκηση πολιτικής και δημόσιας πίεσης, η οποία απαιτεί ε, ταχύ αποτελέσματα από την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν θα πρέπει να παρακάμπτει την κυβέρνηση της ούτε την κοινωνία των πολιτών στη χώρα αυτή. Γνωρίζουμε ότι μεταξύ των εταίρων μας υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που ήδη έχουν πάρει πρωτοβουλίες και που συμμετέχουν στη διανομή της ε, βοήθειας καθώς και την δημιουργία τοπικών δομών. Για παράδειγμα, πολλές τοπικές οργανώσεις προσπαθούν να συγκεντρώσουν κάποια δεδομένη στοιχεία για τους νεκρούς και τους πληγέντες και προκειμένου να δουν ε, επίσης τι μορφή βοήθειας μπορεί να παρασχεθεί στις πληγήσεις οικογένειες. Στο παρελθόν ε, είχαμε πολλά παραδείγματα όπου κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε, δηλαδή δεν συμμετείχαν οι κάτοικοι της ΑΕΤΙΣ. Ε, πολλοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί μπορούν να πιστοποιήσουν την ε, την προσπάθεια των οργανώσεων της ΑΕΤΙΣ να διανύμουν βοήθεια, νερό κλπ. σε εξαιρετικά τις συνθήκες. Το σύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί για την ανοικοδόμηση της χώρας θα πρέπει να συμπεριλάβει την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο επίπεδο της κυβέρνησης, αλλά θα πρέπει επίσης να ληφθεί να ληφθούν υπόψη οι τοπικές αρχές, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τεράστια μετανάστευση αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη προς τις, ε, χώρες, ε, προς τις πόλεις συγγνώμη, στην ενδοχώρα. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί κάτοικοι του Πόρτο Πρένς που εγκαθίστανται σε αυτές τις περιοχές, αλλά εκεί οι κάτοικοι δεν είναι σε θέση να τους βοηθήσουν ούτε να τους παρέχουν την αναγκαία τροφή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια κατεπίγουσα βοήθεια σε αυτά τα κέντρα υποδοχής στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις ε, κατεπίγουσες πρωτοβουλίες για να προωθήσουμε την αξιολόγηση, την ιεράρχηση των αναγκών, όπως ανέφερε και ο κ. Επίτροπος, τόσο όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και ε, την ανοικοδόμηση της χώρας. Γιατί νομίζω ότι είναι ενδεχμένο να ξεκινήσουμε με την ανοικοδόμηση ευθύ αμέσω χωρίς να έχει προηγηθεί ένας απολογισμός και χωρίς ε, επίσης να αξιολογηθούν οι μελλοντικοί κίνδυνοι ε, σεισμών που συνεχίζουν να είναι υπαρκτοί. Ε, στις πρώτες βοήθειες επίσης περιλαμβάνουμε τις ε, τροφές που παράγονται αγοράζονται στην ίδια την αιτία, στο και αν έχουμε συνείδηση ότι αυτή τη στιγμή η επιστημιστική βοήθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αλλά πιστεύουμε ότι μεσοπρόθεσμα και ίσως βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την ε, τοπική γεωργία, την αγροτική οικονομία μπορεί να ανταποκριθεί στις τοπικές ε, ανάγκες με τον πιο δεδειγμένο τρόπο. Όσον αφορά την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια του πληθυσμού, πιστεύουμε ότι τα ακόλουθα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι η κυβέρνηση της ΑΕΤΙΣ που είναι υπεύθυνη για την προστασία των πολιτών της και την εγγύηση των διεθνών πόρων και της διεθνούς βοήθειας και τη συστή κατανομή τους καθώς και την, εφαρμογή, την εγγύηση της εφαρμογής των νόμων από την αστυνομία. Ε, επιθυμούμε να γίνουν προσπάθειες για την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των ε, αστυνομικών, γιατί βεβαίω το σώμα της αστυνομίας έχει απολέσει πολλά από τα μέλη του. Η διεθνής ε, βοήθεια, η διεθνής συνδρομή ε, στη φάση των πρώτων επιχειρήσεων αρρωγής και ανοικοδόμηση, στην πρώτη φάση ανοικοδόμηση της χώρας θα πρέπει να γίνει υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνεργασία με την κυβέρνηση ε, ΑΙΤΙΣ. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί μια πολιτική προστασίας για την, όσον αφορά την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ορισμένες ε, κατηγορίες του πληθυσμού και αυτό ε, και με την ε, συμμετοχή των ε, τοπικών φορέων. Και εδώ γύρεται το ερώτημα κατά πόσο δεν είναι αναγκαίο στο εγγύς μέλλον να αναθεωρήσουμε ενδεχομένως ή να προσαρμόσουμε την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών. Η Αιτή δεν είναι μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο ή σπαράστα από έναν εμφύλιο πόλεμο, αλλά μια χώρα η οποία έχει άμεσα ανάγκη μια στήριξης και κοινωνικής βοήθειας. Όσον αφορά τα διαφορετικά μέτρα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, είναι αναγκαίο να δούμε τι μπορεί να γίνει άμεσα για την ε, ακύρωση του χρέους της, ε, για την απάλληψη του χρέους της χώρας. Ξέρουμε ότι η Ισπανία και η Δημανικανή Δημοκρατία έχουν ξεκινήσει κάποιες ε, δράσεις από την έννοια αυτή. Αλλά αυτή η έκκληση αφορά όχι μόνο τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως είναι η Διεθνής Τράπεζα αλλά ή το Διεθνές Νομισματικό και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά επίσης του δασκούς εταίρους IT όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να ασκήσει πίεση για την ε, απάλληψη του χρέους το ταχύτερο δυνατό. Όσον αφορά την ενίσχυση των κρατικών ε, θεσμών είναι σημαντικό να βοηθηθεί η εθνική κυβέρνηση αλλά επίσης και οι τοπικές αρχές γιατί είναι σημαντικό να αποσυμφορηθεί το Πόρτο Πρένς και να αναζωογονηθεί η επαρχία της χώρας, να μην περιστούμε δηλαδή στην πρωτεύουσα. Ήδη ανέφερα ότι η μετανάστευση προς την Εδωχώρα και τις άλλες ε, πόλεις βρίσκεται υπό εξέλιξη. Τώρα, ένα άλλο σημείο αφορά στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στην ΑΕΤ που μπορούν να βοηθήσουν και θα πρέπει να συμπεριληφθούν ακριβώς στην ε, οργάνωση του κράτους και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, να υποστηριχθεί η κοινωνία των πολιτών της ΑΕΤΗΣ ούτως ώστε να μπορεί να συμμετάσχει ακριβώς σε αυτές τις εργασίες στην υποβολή προτάσεων και σε όλες αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Ε, θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της ανοικοδόμησης επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στις ε, τροτές κοινότητες. Ε, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που υπάρχουν ε, όσον αφορά μια πολύ τρωτή και σεισμοπαθή περιοχή. Ε, όπως είπε ο κ. Ντεχκούχτ, θα πρέπει να σκεφτούμε γύρω από αυτές τις πρωτοβουλίες σχετικά με την ανοικοδόμηση και τα αντισυσμικά μέτρα. Από την άλλη θα πρέπει να εκπονηθούν κάποιες πρωτοβουλίες πρόληψης των κινδύνων που μπορούν να λειτουργήσει σε σχέση με την κυβέρνηση και τοπικούς οργανισμούς. Μετά τις πλημμύρες του 2004 και του 2008 είδαν το φως κάποιες ε, πρωτοβουλίες ε, ορισμένων υπηρεσιών και συστήμα συστήματο προστασίας των πολιτών που λειτουργεί μεν, αλλά που θα πρέπει ασφαλώς να ενισχυθεί και να εξελιχθεί περαιτέρω. Και εδώ προσθέθηκε επίση μια ανάγκη βελτίωσης της ε, τεχνικής της γεωργίας όσον αφορά την ε, μακροπρόθεσμη διαφύλαξη και προστασία των υγεών και την αποφυγή της διάβρωσης, ιδιαίτερα εκεί όπου το έδαφος είναι επικλινές. Αυτή η τεχνική θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διαχείρισης από την τοπική κοινότητα με την στήριξη ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και επίσης του κράτους. Υπό την έννοια αυτή εμείς είμαστε υπέρ της εφαρμογής μιας αγροτικής πολιτικής στην ΑΕΤ με την υποστήριξη της, ε, ε, με τη συνδρομή της διεθνούς βοήθειας. Ε, αυτό αφορά βεβαίως μια βιώσιμη γεωργία και αυτό είναι σημαντικό εάν εφόσον μιλάμε για μια ανόρθωση του κράτους της ΑΕΤ και του πληθυσμού και μάλιστα μακροπρόθεσμα η παραγωγή των τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί με βιώσιμο τρόπο. Οι αγρότες της ΑΕΤ που χρησιμοποιούν μεθόδους που εμείς χρησιμοποιούσαμε στην Ευρώπη των Μεσαίωνα θα πρέπει να βοηθηθούν από πολύ συγκεκριμένε κυβερνητικές αποφάσεις και από πολύ συγκεκριμένε υποδομές. Χρειαζόμαστε λοιπόν τεχνική υποστήριξη για αυτούς. Και θα πρέπει να μπορούν βέβαια να έχουν πρόσβαση και σε πιστώσεις, σε δάνεια. Τώρα, το δικαίωμα ιδιοκτησίας γης και η ασφάλεια ιδιοκτησίας γης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη πέθρου στην ΑΕΤ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολύ μεγάλη ανασφάλεια όσον αφορά την κτήση γης, προβλήματα τα οποία δεν επιτρέπουν στους αγρότες της να προχωρήσουν ε, με τις ε, καλλιέργειές τους. Παρ' όλα αυτά, τελευταία χρόνια είδαμε μια κάποια πρόοδο. Όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις από την κυβέρνηση ενθαρρυντικές πριν από το σεισμό. Ελπίζουμε ότι και στην ενδοχώρα θα μπορέσουν οι αποφάσεις αυτές να εφαρμοστούν. Ένα τελευταίο τώρα σημείο, το οποίο θεωρούμε βέβαια πολύ σημαντικό, πρέπει να αξιολογήσουμε τις πολιτικές και τις συμφωνίες εξωτερικού εμπορίου που υφίστανται με την ΑΕΤ, ανάμεσα στην ΑΕΤ δηλαδή και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στην ΑΕΤ να είναι σε θέση να επιβάλλει εκ νέου φόρους στις εισαγωγές, προκειμένου να ενθαρρύνει την τοπική παραγωγή και προκειμένου να ενθαρρυνθεί κατά αυτόν τον τρόπο όλη η αλυσίδα της παραγωγής τροφίμων, στα πλαίσια της ΑΕΤΗΣ. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν πάλι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρική σχέσης με την ΑΕΤ προκειμένου να ενδυναμωθεί ο γεωργικός τομέας στην ΑΕΤ. Ο τομέα αυτό είναι πολύ σημαντικός για μα. Πρόεδρο, Σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σα αυτή. Το λόγο τώρα έχουν οι βουλευτές για να θέσουν ερωτήσεις στον κύριο Επίτροπο και σε εσά. Το λόγο έχει καταρχάς ο κύριος Μίτσελ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές μας για τις παρουσιάσεις που κάνανε. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, ο οποίος πήγε ο ίδιος στην ΑΕΤ, πήγε και γύρισε πολύ γρήγορα και δεν ξέρω πραγματικά σε τι να αναφερθώ ε, μιλώντας για την ΑΕΤ. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα και την παρουσίαση του Επιτρόπου, καθώς επίσης και την παρουσίαση της εκπροσώπου των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Προφανώς ε, συλληπιτήρια σε όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους και τις οικογένειές τους και ενθαρρυντικά μηνύματα, αν θέλετε, μηνύματα ελπίδας για όλους τους επιζήσαντες. Αν δούμε τώρα τον φάκελο με τα συγκεκριμένα δεδομένα για την ΑΕΤ, πριν τον σεισμό και πριν τον σεισμό έπλητε απίστευτη φτώχεια, απίστευτη ένδια τη χώρα αυτή. Αν δούμε και τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, βλέπουμε ότι το ίμιση του πληθυσμού ζούσε με ένα δολάριο ή κάτω από ένα δολάριο την ημέρα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ποσό του πληθυσμού είχε μόνο δύο δολάρια την ημέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ολόκληρος κατάλογος προβλημάτων για την IT Και είναι πολύ δύσκολο τώρα και με το σεισμό αυτό να συλλάβουμε τη δραματική κατάσταση της χώρας. Να πω καταρχάς ότι χαίρομαι που ο Επίτροπος είπε ότι θα γίνει μία συζήτηση για την οικοδόμηση στον Καναδά, νομίζω ότι είπατε κύριε Επίτροπε. Συμφωνώ μετά όσα είπαν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την ε, εξάλληψη του χρέους, την ακύρωση του χρέους της ε, ITs. 1,2 δισεκατομμύρια ακυρώθηκαν τον Ιούνιο του 2009, αλλά απομένουν ακόμα 800 εκατομμύρια δολάρια. Εκρεμούν ακόμα αυτά ως χρέος και καταλαβαίνετε ότι η IT δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, να αποπληρώσει τέτοιο χρέος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους κατοίκους της IT να κουβαλήσουν και αυτό το βάρος, πέρα από όλα τα προβλήματα που έχουν. Θα ήθελα να επιβεβαιώσει ο Επίτροπο ότι οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια δίδεται αυτή τη στιγμή έχει τη μορφή χορηγία, ε, χορηγίας, επιδότησης και όχι δανείου και πρέπει να πω επίσης ότι μιλήσαμε εδώ, εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε χρησιμοποιώντας τον όρο battle groups, ε, ομάδες ε, μάχης. Νομίζω ότι είναι ατυχής ο όρος αυτός. Μολονότι εμπλέκονται πολλές κοινοτικέ ομάδες δεν καταφέρνουμε να έχουμε μια σημαντική ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε για παράδειγμα όλες τις ειδήσει σε ένα αμερικανικό πλοίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν νοσοκομείο. μονομένα μεμονωμένα κράτη-μέλη έχουν προβεί σε συγκεκριμένε προσπάθειε, το Βέλγιο, η Γαλλία κτλ. και άλλα κράτη θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο. 43 συνολικά νομίζω ότι έχουν συμβάλει. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε μία ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να μην, να μην ονομάζεται αναγκαστικά battle group, ομάδα μάχης που είναι λίγο άγριος επιθετικός όρος, να είναι μία ομάδα παρούσα η οποία θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Νομίζω λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ότι όπως είπε ο Επίτροπος και όπως είπε η κυρία Σόμανς, θα πρέπει να έχουμε κατά νου πώς έχει κατάσταση στην ΑΕΤ και να ενημερωνόμαστε τακτικά. Το, κύριο, το λόγο έχει ο κύριος Ντέβα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Επίτροπο, καθώς επίσης και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για την παραδειγματική δραστηριοποίησή τους στην ΑΕΤ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή τους, ιδίως στο συντονισμό της δικής μας βοήθειας για τη μετώπιση της τραγωδίας αυτής. Θα ήθελα τώρα να πω ότι είμαι στην Επιτροπή αυτή εδώ και δέκα χρόνια και στην περίοδο αυτή έχουμε ασχοληθεί με τσουνάμι στην Ινδονησία, στη Σρι με σεισμού στην Τουρκία, με παλήριες και πλημμύρες ε, στη Μοζαμβίκη, με, κατε... με τυφώνες και κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια μεγάλη φυσική καταστροφή όπως αυτή που έχουμε τώρα στην Αϊτή, φαίνεται ότι ε, ξεκινάμε πάντα από το μηδέν και προσπαθούμε να επανεφεύρουμε τον τροχό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να φαινόμαστε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε τόσο έκπληκτοι από την κατάσταση στην ΑΕΤ. Θα πρέπει ουσιαστικά να αναμένουμε την κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι όντως χρειαζόμαστε πόσιμο νερό, ότι χρειαζόμαστε ιατροφημαρκευτική βοήθεια, χρειαζόμαστε τρόφιμα, χρειαζόμαστε φάρμακα. Χρειαζόμαστε μηχανήματα, γερανούς, ε, ελικόπτερα προκειμένου να καθαρίσουμε τα συντρίμμια. Χρειαζόμαστε κάποιες νέες μορφές ε, στέγασης, χρειαζόμαστε κέντρα φιλοξενίας, χρειαζόμαστε ιατρούς, χρειαζόμαστε νοσοκόμες. Όλα αυτά είναι ευνόητα. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι διαθέσιμα και ένα 80% από τις πολύ μεγάλες ε, καταστροφές που έχουν συμβεί στον κόσμο έχουν συμβεί το πολύ 100 χιλιόμετρα μακριά από την ε, θάλασσα. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαν εδώ πέρα να είχαν προβληφθεί οι απαραίτητε δομέ που θα επέτρεπαν τη μεταφορά των ανθρώπων στην εδωχώρα και θα είχαν σωθεί κατά αυτόν τον τρόπο πάρα πολλέ ζωέ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από κάποιο κράτος μέλος να παρέχει τα παρέτα ελικόπτερα τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Όταν για παράδειγμα είχαμε την καταστροφή στην ε, Μοζαμβίκη Είχα παρενέβω ίδιο ίδιος προκειμένου να ζητήσω από κράτη-μέλη να παρέχουν τι απαραίτητες δυνάμεις, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον πλοίο αυτό, το οποίο τελεί χρέη νοσοκομείου, το ιατρικό προσωπικό το οποίο είναι μέσα στο πλοίο αυτό, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μηχανήματα και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι παρόντες προκειμένου να βοηθήσουμε την κατάσταση στην Αιτή για παράδειγμα, στο τσουνάμι για πάρα πολλούς μήνες, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εκεί, έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το τοπικό αεροδρόμιο και δεν καταφέρναμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να φύγει από την περιοχή και προφανώς είχε είχε... υπήρχε φοβερή κίνηση και συμφόρηση στο αεροδρόμιο αυτό. Προφανώς δεν γινότανε να εξυπηρετήσει το αεροδρόμιο αυτό όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχαν τα απαραίτητα αυτά μέσα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, ειδικά διαμορφωμένα, τα οποία μπορούσαν να μεταφέρουν τον κόσμο. Κατά αυτόν τον τρόπο, αν είχαμε χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά και στην ΑΕΤ, θα μπορούσαμε να είχαμε βοηθήσει τον κόσμο άμεσα. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχουν αυτή την υποδομή στι άλλε περιοχέ του κόσμου που πλήττονται αυτή τη στιγμή από φυσικέ καταστροφέ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο χρόνος ομιλίας πρέπει να περιοριστεί στα δύο λεπτά. Κύριε Γκερέρο, έχετε τον λόγο. Ήθελα να ε, επαναλάβω και εγώ τα συγχαρτήρια προς τους μη κυβερνητικού οργανισμούς και τον Επίτροπο για το έργο του στην ΑΕΤ και θα ήθελα επίσης να εκφράσω και τα δικά μου συλλεπιτήρια για τους χιλιάδες χιλιάδων ε, κατοίκων της έτη τους. Θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή μου σε ένα από τα τρία στοιχεία στα οποία ανέφερε και ο κ. Επίτροπος και αφορά την ε, ανοικοδόμηση ενός κράτους που να λειτουργεί εύρυθμα. Η ΑΕΤ είναι μια χώρα σε ιδιαίτερα αξιοθρύνητη κατάσταση. Ακόμα και πριν από την καταστροφή ήταν μια χώρα εξαιρετικής ένδυας. Ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα και επίσης μια χώρα με κακές σχέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες. Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν, πρόκειται για ένα αχροκοπημένο κράτος και γι' αυτό πολλοί, ακόμα και κάτοικοι της ΑΕΤ, λένε τώρα ότι δεν θα πρέπει να ανοικοδομηθεί η ΑΕΤ, θα πρέπει να οικοδομηθεί η ΑΕΤ και για να οικοδομηθεί η ΑΕΤ θα πρέπει να λυθεί ε, το πρόβλημα της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας ε, και θα πρέπει να εξελιχθούν προς μία μορφή μετάβασης. Και νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαρματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της χώρας, στην οικοδόμηση μιας χρηστής διακυβέρνησης, δηλαδή πρικοδοτώντας τη νέα ΑΕΤ με εκείνες τις ε, πολιτικές ε, δομές που απουσίαζαν στο παρελθόν, που οδήγησαν στην αποτυχία και βρίσκονται τις απαρχές των ε, τρομακτικών προβλημάτων που υπήρχαν ήδη πριν από την καταστροφή του σεισμού. Κύριε Γκέρνς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία σημεία. Πρώτον, νομίζω ότι απαιτείται μια έκθεση αξιολόγησης της κατάστασης και της προστιθέμενης αξίας την οποία μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε για το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο χρόνο, γιατί σε λίγες μέρες κανένας δεν θα ασχολείται με την IT και εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες για την προσπάθεια α, ανόρθωσης της χώρας. Εγώ δεν είμαι υπέρ της κατάργησης του χρέους γιατί δεν είμαι υπέρ των <clears throat> δανείων που δίδονται στις υποανάπτυξη χώρες. Αν έχουν δοθεί τα χρήματα, θα πρέπει να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της απόσβεσης. Δεν θα πρέπει εμείς να αποεπευθυνοποιήσουμε αυτούς οι οποίοι δανείζονται χρήματα. Αν δεν ήταν η βοήθεια που δώσαμε μέχρι τώρα ικανοποιητική, δεν θα πρέπει να τους υποχρεώσουν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο αν απέτυχε. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα τύπου EU Fast, το οποίο θα έχει αποκλειστικά ανθρωπιστικό και μη στρατιωτικό χαρακτήρα, μόνιμο όμως, θα κινητοποιείται ο μηχανισμός αυτός κάτω από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα, θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα συνεργάζεται με τρίτες χώρες, θα είναι διαθέσιμη η δύναμη αυτή για την συνεργασία της στην αγαστή με ε, τα Ηνωμένα Έθνη και με τους αντίστοιχους μηχανισμούς των κρατών μελών. Θα πρέπει να ανοίξει ένας κατάλογος, να καταρτιστεί ένας κατάλογος των δυνατοτήτων που θα έχει ανάγκη αυτό το EU Fast και θα πρέπει να ενημερώνεται ο κατάλογος αυτός συνεχώς. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα, ένα σύστημα το οποίο επαναλαμβάνω θα πρέπει να έχει μη στρατιωτικό χαρακτήρα, γιατί υπάρχουν δυνατότητες στο στρατιωτικό δομέα οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν κάτι τέτοιο είναι αναπαραίτητο. Αλλά χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους μέσα στρατιωτικά δεν σημαίνει ότι μετατρέπουμε τη δράση μας από μη στρατιωτική σε στρατιωτική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσπάθεια. Κυρία Λάντφορντ, δύο λεπτά. Δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο πάντως. Ξέρω ότι ο κύριος Ντίβα παρακολουθεί τα θέματα αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο να μου πει ποιες είναι οι προοπτικές για μία θα έλεγα ομάδα ευρωπαϊκή ή το Eurofast ή το Euro κάτι εν πάση περιπτώσει κάτι το οποίο να παρεμβαίνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Συμφωνώ με αυτούς που μίλησαν προηγουμένως, το θέμα δεν είναι μόνο της εικόνας της Ένωσης, κάτι το οποίο δεν πρέπει να υποτιμάμε, αλλά το θέμα είναι κυρίως θέμα αποτελεσματικότητας. Έχω μια μικρή σύγχυση γιατί ο κύριος το κρίνει θετικά γενικά τον τρόπο με τον οποίο καλύφθηκαν οι ανάγκες και αυτό διαφέρει από τις εκθέσεις οι οποίες παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης όταν ο κύριος Ντίβα είπε ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να συντονίσει κανείς τα κράτη-μέλη, έκανε μια μικρή γκριμάτσα ο κύριος Ντεγκούχτ. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα δεν πετύχαμε μια τέτοια ενιαία μορφή ευρωπαϊκής αντίδρασης ή προσπάθειας. Υπάρχουν από εδώ και πέρα καλύτερες προοπτικές. Δεν ξέρω τι ακριβώς δίνει δυνατότητες, ποιες ακριβώς δυνατότητες δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας, δεν τον ξέρω τον τομέα εγώ προσωπικά καλά, αλλά μήπως το περιβάλλον είναι καλύτερο για τη δημιουργία μια συντονισμένης ευρωπαϊκής μορφής αντίδρασης σε τέτοιου είδους καταστάσεις, όπου από πριν θα ξέρουμε το ποιος θα κάνει τι. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, λέει η κυρία Ζολή, 10 δευτερόλεπτα για τις Το θέμα είναι να βοηθήσουμε και την αγορά τροφίμων τοπικά έτσι ώστε να βοηθήσουμε να ξεκινήσει ξανά και η γεωργία η τοπική. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Ντεχούχτ. Όλοι βιώσατε αυτή την τραγωδία και άκουσα να λέτε ότι η Ευρώπη θα είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ικανοποιεί. Η Αιτία είναι επίσης μια χώρα στην οποία η βία εις βάρος των γυναικών και η σεξουαλική βία έχει τρομερές διαστάσεις. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι με αυτό το σεισμό φυσικά τα πράγματα χειροτερεύουν γιατί πολλές γυναίκες αναγκάζονται να εκδίδονται για να έχουν καθαρό νερό μόνο. Και υφίστανται επίσης και αυξήσεις στα επίπεδα συζυγικής βίας. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια αυτής της κατάστασης στα πλαίσια της προσπάθειας αποκατάστασης θα λάβει υπόψη την θέση την ευάλωτη των γυναικών και των κοριτσιών, γιατί έχουν συγκεκριμένες ανάγκες σε διάφορους τομείς, ε, όπως σε επίπεδο μέτρων αντισύλληψης ε, ε, και τα λοιπά. Ποιο είναι το μέλλον του στην Αιτή, Κυρία Στρίφλερ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγκούχτο για τις πολύτιμες ε, πληροφορίες του. Θα προτείνω μία συνάντηση με τους συντονιστές να δούμε πώς θα είμαστε αναπόσπαστο τμήμα αυτής της προσπάθειας ανοικοδόμησης. Ανακοινώσατε μια νέα παρέμβαση ανθρωπιστική 19 εκατομμυρίων ευρώ για την κατεπίγουσα βοήθεια ποιοι είναι οι άξονες αυτής της κατά προτεραιότητα λήψης απόφασης καλύπτεται και άλλες πόλεις που θίγονται εκτός από την πρωτεύουσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμα το 2007 ζήτησε τη δημιουργία μιας ειδική ομάδας εργασίας στο εσωτερικό του Συμβουλίου έτσι ώστε να ακολουθηθούν κοινέ μέθοδοι για τη διευκόλυνση μεθόδων άμεσης ανταπόκρισης σε τέτοιες καταστροφές κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να εμβαθύνουμε τη συζήτησή μας για την πολιτική που θα ακολουθούμε στην ανθρωπιστική βοήθεια. Δημιουργήθηκε στις 1η Ιανουαρίου του 2009 και μια ομάδα εργασίας. Τι ρόλο έχει αυτή η ομάδα η ΚΟΑΦΑ στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού στην ΑΕΤΗ. Ο κύριος Στάις, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κάρελ Ντεγκούχτο για μια σαφή ε, παρέμβαση. Ευχαριστώ επίσης και την κυρία Σόμαν. Ε, κάποια από τις ερωτήσεις που έχω να θέσω τις έχουν θέσει και άλλοι συνομιλητές. Το θέμα είναι ε, για αυτή την πιθανή ε, δύναμη σε εισαγωγικά το Eurofast. Υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για τη δημιουργία της σήμερα από ό,τι πριν το σεισμό. Μιλώντας για τις ΜΚΟ, δεύτερη ερώτηση. Μιλάμε για εμπορική πολιτική, για εταιρικές σχέσεις που πάρα πολύ συχνά δεν είναι ευνοϊκές ε, ε, για τους ε, πληθυσμούς. Μήπως εκεί μπορεί να δει κάποια βήματα προόδου εύκολα να γίνουν στο μέλλον ο κύριος Δεγκούχτ. Έχει ζητήσει επίσης το λόγο η κυρία Σάνκτη. Εννοεί την κυρία Τσανίκη η πρόεδρος. Ο σεισμός αυτός μας έχει πραγματι όλους συντρίψει και όλοι θέλουμε κάπως να βοηθήσουμε και η Ιταλία ήταν μια από τις χώρες η οποία ξεκίνησε με 200 γιατρούς και ένα νοσοκομείο εκστρατείας, στείλαμε αεροπλάνα με φάρμακα κτλ. Θα ήθελα να μην αναφερθώ σε αυτό όμως, να θέσω το εξής. Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει σαν γυναίκα, μητέρα και γιαγιά είναι η εικόνα του να βλέπουμε παιδιά τα οποία έχουν χαθεί, είναι μόνα τους πια και υφίστανται χρήσης, έχουν γίνει σκλάβοι τα παιδιά αυτά, ακούσαμε φρικτά πράγματα. Για αυτά τα παιδιά δεν μιλάει κανείς πια. Τι γίνεται για αυτά τα παιδιά, γίνεται κάτι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά είναι τρομερό. Δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά τα οποία έχουν χαθεί, είναι αγνοούμενα τώρα. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά καλό είναι να τεθεί το θέμα της τύχης των παιδιών αυτών. Ο κύριος Ντεγκούχτ. Για πέντε λεπτά παρακαλώ. Προσπαθήσω πρόεδρε. Ο κύριος Μίτσελ είπε ότι ένα 77% του Πόρτο Πράνς έχει καταστραφεί. Δεν ισχύει αυτό. 20% του Πόρτο Πράνς έχει καταστραφεί θα έλεγα. Και επίσης έχουμε πόλεις όπως η Λεογκάν, Μέλ και στις οποίες έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ περισσότερο πολλές φορές από ό,τι στο Πορτοπράνς. Το Πόρτο Πράντς βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη πόλη και όπως εξήγησα έχετε ορισμένες περιοχές που έχουν καταστραφεί εντελώς ενώ άλλες δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα σχετικά γειτονικές περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα. Δρόμοι που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την οποία βρίσκονταν πριν από το σεισμό. Και αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θεωρώ λοιπόν ότι να λέμε ότι ένα 70% του πορτοπράσι καταστραφή δεν είναι σωστό. Μα αυτό λέγεται στην έκθεση που μου έχει δοθεί από μη κυβερνητικέ οργανώσει. 77% των κτηρίων έχει καταστραφεί. Αυτό λέγεται. Απάντηση του Επιτρόπου δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πήγα επιτόπου Πήγα σε πολλά μέρη μέσα στην πόλη την είδα από διάφορες πλευρές αν θέλετε. Έφτασα, έφυγα από την πόλη, την είδα και από ελικόπτερο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα 20-25% το πολύ της πόλης έχει καταστραφεί, που σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Τρία με τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπων ζουν στο πορτο Πράντς, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι 70-77% του πορτο Πράντς έχει καταστραφεί. Τουλάχιστον εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο και είμαι εδώ για να σας πω ότι είδα. Αναφερθήκατε στα δάνεια στη συνέχεια. Όλα τα χρήματα που διατίθενται αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση της ΑΕΤ και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και για την ΟΕΕ είναι επιχορηγήσει ουσιαστικά. Είναι επιδοτήσει, είναι, δεν είναι δάνεια, δεν, έχει, δεν θα, υπήρχε, θα ήταν παράλογο αυτή τη στιγμή να δώσουμε δάνεια. Σε καμία περίπτωση θα κάνουμε κάτι τέτοιο, θα ήταν παράλογο. Πολλέ ερωτήσει ε, ακούστηκαν για το EU Fast, για την εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μελλοντικέ προοπτικέ παρεμβασή μα. Καταρχά πρέπει να σα πω ότι με την επόμενη Επιτροπή η ανθρωπιστική βοήθεια και η προστασία των πολιτών θα αποτελέσουν αντικείμενο του ίδιου χαρτοφυλακίου ενός επιτρόπου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πιστεύω. Και μην ξεχνάμε ότι η προστασία των πολιτών αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο συντονιστικός μηχανισμός που έχουμε υιοθετήσει, ο MIC, θα ανήκει πλέον στο ίδιο χαρτοφυλάκιο με την ανθρωπιστική βοήθεια και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου. Επίσης, στην συνθήκη της Λισαβόνας τα πράγματα είναι πολύ πιο σαφή και συγκεκριμένα όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σαφήνεια αυτή προκειμένου να υποβάλουμε περισσότερες προτάσεις και επίσης στη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει σαφής ρήτρα αλληλεγγύης, πράγμα το οποίο δεν είχαμε με προηγούμενες συνθήκες. Και σε περίπτωση μια τέτοια καταστροφή θα μπορούσε αργά ή γρήγορα να συμβεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου και ήδη η συνθήκη προβλέπει εργασία των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα αυτό. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω τη ΕΚΟ, μια υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λειτουργεί πολύ καλά. Έχουμε την MIC που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του κύριου Δήμα και από ό,τι μπορούμε να πούμε έχει λειτουργήσει πολύ καλά η MIC στην κρίση αυτή, κινητοποιήθηκε πολύ γρήγορα και ουσιαστικά αυτό που προβλέπεται στην MIC είναι ότι κινητοποιούνται ικανότητες από τα κράτη-μέλη. Μπορεί ο συντονισμό να μην ήταν πολύ καλός και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε έναν στονιστικό μηχανισμό, τον EUCO, που στόχος του είναι να συγκεντρώσει τις στρατιωτικές δυνάμεις ικανότητες από τα κράτη-μέλη που όπως είπατε βέβαια και πολλοί, αυτό δεν σημαίνει ότι προχωρούν σε στρατιωτικές συναγκαστικά επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι η παρέμβαση του στρατού είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη σε τέτοιες κρίσεις. Αυτούς λοιπόν τους μηχανισμούς έχουμε, οι οποίοι λειτουργήσαν πολύ καλά και τουλάχιστον πολύ καλύτερα από ό,τι στο τσουνάμι που είχαμε στο παρελθόν. Μπορούμε να πούμε ότι οι φυστάμενοι μηχανισμοί όσοι έχουν αυτή τη στιγμή λειτουργήσαν πολύ καλά, σαφώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν, σαφώς τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν και για αυτό το λόγο θα έχω πολύ σοβαρές συζητήσεις με τον άνθρωπο που θα αναλάβει το δικό μου το χαρτοφυλάκιο προκειμένου να δούμε πώς θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα τροτά στοιχεία του μηχανισμού. Η ορατότητα εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με τη δυνατότητα σωστής λειτουργίας επιτόπου και με την ε, δυνατότητα που θα έχουμε να συνδυάσουμε πολλές ικανότητες, όπως είπατε και εσείς κύριε Ντέβα, δηλαδή να έχουμε πλοία πολυχρηστικά, τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν πάρα πολλές καταστάσεις. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητο συντανισμό, η απαραίτητη οργάνωση προκειμένου ένα τέτοιο πλοίο να είναι παρόν όταν πρέπει να είναι παρόν. Ενδεχομένω θα μπορούσατε εσεί να κάνετε μία πρόταση για την ε, απαραίτητη χρηματοδότηση και οργάνωση για τη χρησιμοποίηση των μηχανισμών. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να στηθεί ένα τέτοιο μηχανισμό. προκειμένου να κινητοποιηθούν όλε τι δυνατότητε που χρειάζονται, όλε οι ικανότητε που χρειάζονται για την αντιμετώπιση μια κρίση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μα απασχολήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου να γίνει η συζήτηση αυτή και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ακούστηκε και μία πρόταση σήμερα στο Συμβούλιο για μία ομάδα θελοντών Πολύ καλή πρόταση. Και ανάλογη πρόταση θα μπορούσαμε εμείς να υποβάλουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά το να θεωρούμε ότι μπορούμε με θελοντές και μόνο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε περιπτώσεις όπως η IT είναι κάπως ε, υπερβολικό. Κάθε φορά που προκύπτουν καταστροφέ στην αυτή τη αιτή, χρειαζόμαστε πραγματικά ειδικού, ειδήμονε στον τομέα του, ειδικευμένα άτομα. Αυτό χρειαζόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί οι δήμονες ειδικοί μπορούν πραγματικά να οργανωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, ε, έχουν εκπαιδευτεί για να εργάζονται ακριβώς σε δύσκολα, δυσχερή περιβάλλοντα. Βέβαια, δεν τα λέω αυτά για να σας πω ότι τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά. Οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας λειτουργούν σωστά στην ΑΕΤ, όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά τα πράγματα λειτουργούν σωστά. Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ορατότητα, αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης, θα έλεγα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αποκλειστικά. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι από όλα τα κράτη-μέλη πηγαίνουν προωθώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε όντω θα είχαμε πολύ μεγάλη ορατότητα και θα βελτιωνόταν η εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω. Ε, ας το παραδεχτούμε, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν, αν θέλετε, τη σημαία της Ευρωπαϊκή Ένωση και δίπλα στη σημαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν και τη δικιά του σημαία αλλά τελικά τα κράτη-μέλη δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βοηθούν, που μπορούν και βοηθούν, αλλά ουσιαστικά δεν προωθούν την ε, εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθούν περισσότερο, αν θέλετε, την εικόνα της σημαία του συγκεκριμένου κράτους. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στο θέμα της βελτίωσης εικόνας Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αποκατάσταση, την ανοικοδόμηση, την οικοδόμηση, την ανοικοδόμηση. Κύριε Γκέρεν, σίγουρα η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει. Και σίγουρα θα μιλήσουμε για οικοδόμηση. Μέσω της ανοικοδόμησης όμως. Τον οικοδομήσουμε όμως ε, μία χώρα, το να δημιουργήσουμε θεσμούς, είναι πολύ πιο εύκολο στο χαρτί θεωρητικά από ότι στην πράξη. Και σίγουρα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα αν είχαμε όμως την πολιτική ηλίτ, την κοινωνία των πολιτών επί τόπου διαθέσιμη. Αν πραγματικά δηλαδή έχετε τις αρχές, τις τοπικές, τις εθνικές διαθέσιμες για να τις υποστηρίξουν. Διαφορετικά, αν απουσιάζει η υποστήριξη αυτή, αν απουσιάζει αυτή η συνεργασία, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο αποβάλαμε μία πρόταση προκειμένου να ανοικοδομήσουμε το κράτος αυτό, την IT, με τη συμμετοχή όμως του ίδιου του κράτους, προκειμένου να μπορούν και οι ίδιοι θύντες να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας τους. Σίγουρα όμως αυτό δεν είναι εύκολο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Αύριο το πρωί θα σας στείλω και μια γραπτή έκθεση με όλα αυτά τα στοιχεία είναι έτοιμη. Θα σας τη στείλουμε μέσω της γραμματείας και εσείς μπορείτε να τη δώσετε συνέχεια στους συναδέλφους σας, στα μέλη της Επιτροπής σας, κυρία Ζολή. Η Σάρα Λάτφορτ. να αγοράσουν οι κάτοικοι τα τρόφιμα, δυνατότητα αγοράς των τροφίμων επιτόπου. Σίγουρα αυτό θα πρέπει να είναι δυνατό, αλλά αυτό σημαίνει στον ουσία ότι θα πρέπει να αγοράζει κανείς τα τρόφιμα μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα δικά μας αποθέματα. Το να αγοράζει κανείς από τις Ηνωμένε Πολιτείες γάλα, για παράδειγμα, σηκώνει γάλακτος, σίγουρα αυτό μπορεί να γίνει, αλλά ας δούμε και τα αποθέματα που έχουμε επιτόπου. Προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα στη συνέχεια για την προστασία των κοριτσιών και των γυναικών. Είμαστε σε επαφή με τη UNICEF, η οποία έχει την συγκεκριμένη αυτή εντολή προστασίας των γυναικών δηλαδή. Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα ορφανά στην τα παιδιά που έχουν μείνει ορφανά και προσπαθούμε να συλλέγουμε και πληροφορίες για την εμπορία παιδιών και να ξέρουμε τελικά πραγματικά πώς έχει η κατάσταση, τι είναι αλήθεια και τι όχι. Να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή να οριοθετήσουμε σωστά το πρόβλημα προκειμένου να υποστηρίξουμε και εμείς τις δράσεις των κρατών μελών και τις δράσεις της UNICEF οποιαδήποτε μορφή απαιτηθεί τελικά για τις δράσεις αυτές, οποιαδήποτε μορφή και αν πάρουν. Ασχολούμεθα και με τις άλλες πόλεις, με το Λεογκάν, αναφέρθηκα σε αυτό. Αναφέρθηκα στις πόλεις εκείνες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο, αλλά υπάρχουν και μικρότερες ε, πόλεις. Το Λεογκάν έχει 105.000 κατοίκους περίπου. Υπάρχουν όμως και ε, άλλες πόλεις με λιγότερους κατοίκους που έχουν πληγεί. Σαφώς η μεγαλύτερη καταστροφή αυτή τη στιγμή είναι ορατή στο Port au Prince. Αλλά έχουμε εκθέσεις μας δείχνουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια έχει οργανωθεί και στις άλλες πόλεις. Ε, ε, ε, θέστε κάποια ερωτήματα και στα Ολλανδικά. Το εμπόριο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην όλη διαδικασία νοικοδόμησης. Στο παρελθόν είχα αναφερθεί στον τρόπο εκείνο με την οποία θα καταφέρναμε να αντιμετωπίσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια πιο αποτελεσματικά, πιο καλά διαρθρωμένα. Νομίζω ότι γενικότερα αναφερόμενο σε μια περιοχή σαν την Καραϊβική θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εμπόριο. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεργασία όσον αφορά το εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντική μεταξύ των δύο κρατών που βρίσκονται πάνω στο νησί της Αιτής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σόμανς, προκειμένου να απαντήσει και αυτή στις ερωτήσεις που της ετέθησαν. Ναι, ε, θεωρώ ότι πρόκειται κυρίως για δύο ερωτήσεις. Οπότε μία όταν λέγαμε ότι θα πρέπει να αγοράζονται οι τροφές επιτόπου, ε, το θέμα δεν είναι να αγοράζονται τα τρόφιμα, αλλά να δίδεται η δυνατότητα στους εγχώριους παραγωγούς, στους αγρότες της ΑΕΤ να βρουν μια αγορά σε τοπικό επίπεδο και έτσι να μπορούν να παραγάγουν για να έχουν κάποια έσοδα, δηλαδή να ενισχυθεί η τοπική αγροτική οικονομία και με τον τρόπο αυτό να ενισχυθεί και η οικονομία και η κατάσταση των μικρών χωρικών που βρίσκονται στην εδώ και που είχαν εγκαταλείψει τη γεωργία σε μεγάλο βαθμό γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή ρυζιού που πωλείται στην αγορά λιγότερο ακριβά από την εχώρια παραγωγή των αγροτών, της, των γεωργών της ΑΕΤΙΣ. Αυτή είναι μια εξέλιξη που έχει διαπιστωθεί τα τελευταία 15 έτη, δηλαδή ότι η χώρια παραγωγή μειώθηκε κατά πολύ λόγω του ανταγωνισμού των εξωτερικών εισαγωγών. Τώρα, ίσως μια σύνομη απάντηση όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών και αυτά που θα απογίνουν στην ΑΕΤ της ε, βίας που ε, υπάρχει στη χώρα, που κυβερνάει στη χώρα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες επίσης όσον αφορά τη βία τις τελευταίες ημέρες ε, την οποία φαίνεται ότι έχουν υπερβάλει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλες αυτές οι εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου και τα διάφορα τηλεοπτικά κανάλια. Γνωρίζουμε ότι ένας τομέας που λειτουργεί πολύ καλά στην ΑΕΤ είναι ακριβώς η οργάνωση γυναικών και γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων πάντοτε λειτουργήσε καλά στην ΑΕΤ, στην όχι μόνο σε αφορά τη βία κατά των γυναικών, αλλά μέσα στο Υπουργείο αυτού υπήρξαν κάποιες δράσεις στο, τομέα της, στο πρόληψης και της ενημέρωσης για το AIDS. Δυστυχώς μάθαμε ότι τρεις από τις ε, ε, γυναίκες αυτές που ήταν πολύ σημαντικές στο γυναικείο κίνημα έχασαν τη ζωή τους στην του σεισμού. Όσον αφορά τη βοήθεια και όχι μόνο την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και μελλοντικά τη μορφή που θα προσλάβει αυτή η βοήθεια. Θα θέλαμε να υποβάλουμε την πρόταση, μάλλον να υπογραμμίσουμε την πρόταση που έγινε από τον κύριο Κούχτ. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε την αύξηση του συντονισμού μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή κάθε χώρα να μην αποστέλει τις ε, διάφορες ομάδες βοήθειας επιτόπου, αλλά να υπάρχει εκ των προτέρων ένα συντονισμός για την αποστολή βοήθειας και η κάθε χώρα να ειδικεύεται σε ένα τομέα για να μην ε, γίνεται αυτή η ad hoc προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε πολύ και τους δύο μιλητές που μας ενημέρωσαν τώρα το μόνο μας απομένει να δούμε πότε θα είναι η προσοχή μας συνεδρίαση. Θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες την Τετάρτη στις 3 Φεβρουαρίου για την ακρόαση της κυρίας υποψηφίου επιτρόπου Γεωργίευα Ζωζίευα από τις 12.30 έως τις 3.30 το μεσημέρι την 5η 4 Φεβρουαρίου από τις 9 έως τις 12.30 και στις 23 Φεβρουαρίου από τις 3 ως τις